good afternoon everyone, ladies and gentlemen. It's 10 past. Καλό σα απόγευμα, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε. Είναι και 3 και 10. Καλώ ορίσατε όλοι και περνάμε απευθεία στο σημείο υπαριθμό υπαρθμό τη μισή διάταξη, έγκριση τη ημερήσια. Εάν δεν έχετε σχόλια μπορούμε να την εγκρίνουμε λοιπόν. Πολύ ωραία. Υπαριθμών 2. ανακοινώσει του Προέδρου δεν υπάρχουν από την πλευρά μου, οπότε περνάμε στο σημείο 3. Ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση σχετικά με την κατάσταση στι Μαλδίβε. Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Ντίπ Μακρίστα, ε, που είναι υπεύθυνο για το Αφγανιστάν, Πακιστάν, Σρι Λάνκα ε, και Μαλδίβε και Μπαγκλαντέ. Χαίρομαι που βρίσκεστε εδώ μαζί μα, ε, έστω και τελευταία στιγμή που σα καλέσαμε. από την ομάδα GUE NGL ήρθαν σε επαφή μαζί μου και μου ζήτησαν να μπει το θέμα των Μαλδιβών στην ημερήσια διάταξη και θέλω να, θέλω σε ευχαριστήσω γι' αυτό. Φαντάζομαι ότι όλοι συμφωνούμε ότι οι εξελίξεις ε, στις Μαλδίβες έχουν επιδεινωθεί. Υπάρχει έλλειψη σεβασμού στην ε, ειρηνική έκφραση αντιπολίτευσης. Υπάρχει σαν υψηλός αριθμός επίσης ε, ξενομαχητών που πάνε στον ISIS, δεν υπάρχει σεβασμό των θεμελιών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Πρόσφατα ε, ε, είχαμε μια δολοφονία σε σχέση με το μέτωπο Γιασμίν Ρασίντ και αυτό ήρθε να επιδεινώσει τα πράγματα. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση θα ήθελα να σας ζητήσω κύριε Κρίσλα να μας κάνετε μια σύντομη παρουσίαση της κατάστασης στις Μαλδίβες και στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον κύριο Κρίσλερ αν δεν έχετε αντίρρηση. Λοιπόν, έχουμε χρόνο έως τις και μισή για αυτό το θέμα, οπότε <laughs> παρακαλώ να είστε όσο γίνεται πιο Σε Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Εκτιμώ ιδιαίτερα τη δυνατότητα που μου δίνεται να ανταλλάξουμε απόψεις για την κατάσταση στις Μαλδίβες με την Επιτροπή σας. Ε, να σας πω καταρχήν ότι οι Μαλδίβες το 2008 ε, ήταν πολλά υποσχόμενη χώρα, μια, σε μια φάση μετάβασης, ε, εκδημοκρατισμού από ένα αυταρχικό καθεστώς σε ένα πολυκομματικό. Ε, ο πρόεδρος Τζαμέν όμως το 2013 έχασε την εξουσία και έκτοτε η κατάσταση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες στη χώρα είναι εξαιρετικά ανησυχητικά. Πολλοί ηγέτες αντιπολίτευσης είναι στη φυλακή, είναι περιορισμένοι από η δραστηριότητά τους και αυτό οφείλεται ε, στον εξαιρετικά αμφιλεγόμενο αντιτρομοκρατικό νόμο. Επίσης υπάρχει μείωση του δικαιώματος έκφρασης και του δικαιώματος ε, συνάθρησης και βεβαίως κάποιοι δημοσιογράφοι και ακτιβιστές δέχονται απειλές και παρενοχλήσεις. Υπάρχει και απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της, ε, των Μαλδιβών. Ε, σύμφωνα με αυτή την απόφαση, το δικαστήριο θα έχει το δικαίωμα να καθορίσει ε, την, ε, τον, τον ομότυπο των αποφασών του Κοινοβουλίου. Περιορίζει δηλαδή το ρόλο του Κοινοβουλίου και ουσιαστικά του αφαιρεί εξουσίες. Ένα άλλο πεδίο ανησυχίας έχει να κάνει με το μορατόριο που έχει δημιουργηθεί de facto για την θανατική ποινή. Υπήρχε ένα μορατόριο για πολύ καιρό σε ό,τι αφορά την θανατική ποινή, όμως η πρόσφατη κυβέρνηση δημοσίως έχει δεσμευθεί ότι θα επαναφέρει τη θανατική ποινή και τις εκτελέσεις. Για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων τώρα, αναγνωρίζουμε ότι έχουν γίνει προσπάθειες από την κυβέρνηση για να βελτιωθεί η θεσμική, το θεσμικό πλαίσιο της χώρας στο ζήτημα αυτό, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει, ε, υπάρχουν σημαντικά, ε, σημαντικές εκδηλώσεις βίας, ε, και κατάχρησης, ε, καταπίεσης των γυναικών. Σε ό,τι αφορά τη βία και τον εξτρεμισμό τώρα που είναι πολύ προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ε, έγινε μια τροπολογία του αντιτρομοκρατικού νόμου ε, του 2015 που καθιστά έγκλημα και παράνομο κάποιος να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε ομάδα που ενδέχεται με τρομοκρατικές επιθέσεις. Όμως περίπου, έχουμε περίπου μισό εκατομμύριο τουρίστες ε, προς τις Μαλδίβες και θέλουμε να συνεργαστούμε ε, σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα μαζί τους. Κύριε Πρόεδρε, αναφερθήκατε ήδη στην περίπτωση της δολοφονίας, της βίας δολοφονίας του blogger από τις Μαλδίβες του κ. Τζαμίν Ρασίδ. Ήταν ένας blogger λοιπόν που δολοφονήθηκε τον Απρίλιο του 2017. Ο κ. Ρασίδ ήταν στόχος πολλών απειλών ε, για τη ζωή τους, για εσωτερικά τους, εσωτερικά του μηνύματα για πολιτικοκοινωνικά ζητήματα, καθώς ε, και διότι ήταν υπέρ ενός κοσμικού κράτους. Η, η αστυνομία των Μαλδιβών έχει συλλάβει μια σειρά από υπόπτους που ενδεχομένως να πραγματοποίησαν το έγκλημα αυτό. Όλα τα ζητήματα στα οποία αναφέρθηκα και ακόμα μερικά τέθηκαν στην τρίτη ετήσια ε, συνάντηση πολιτικού διαλόγου μεταξύ Ευρωπαϊκής και Μαλδίβων που ε, έγινε υπό την αιγίδα του, του Υπουργού Εξωτερικών στις 31 Μαΐου. Πλέον οι Μαλδίβες δεν χαίρουν ενίσχυση για την ανάπτυξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν εκπροσωπείται στις Μαλδίβες. Όμως θεωρούμε ότι υπάρχουν δυνατότητες διαλόγου και συνεργασίας με την κυβέρνηση των Μαλδίβων και θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες από τις δυνατότητες αυτές από δικής μας πλευράς τουλάχιστον. Καταρχήν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει ε, την επιρροή της για να πιέσει την κυβέρνηση των Μαλδιβών να αξιολογήσει ε, την απειλή της ε, σπαστικοποίησης των νησί. Θα μπορούσε να βοηθήσει το κέντρο το δημοκρατικό της χώρας, με δημιουργία δυνατοτήτων για την αντιμετώπιση ε, των ε, εξτρεμιστικών ακραίων βίων ε, αφηγήσεων και λόγου. Θα γίνει και μια διάσκεψη αντιτρομοκρατική στις Μαλδίβες πριν από το τέλος του έτους και ο συντονιστής του αντιτρομοκρατικού γραφείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Σίλ Τεκέρκοφ, θα συμμετάσχει. Επίσης πρέπει να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις σε ό,τι αφορά το εκλογικό σύστημα και τι εκλογέ θα πρέπει να υπάρξει ομάδα παρατηρητών από την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε οι επόμενε εκλογέ να είναι αξιόπιστε διαφανεί και συμπεριληπτικές. Οι προεδρικέ εκλογέ θα λάβουν χώρα στις 2000, το, το, το 2018 και θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση να στείλει παρατηρητέ Η κυβέρνηση των Μαλδίβων έχει επίση καλέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει μια ενδιάμεση αξιολόγηση μετά τις προεδρικές εκλογές του 2013 όπου επίσης υπήρχαν παρατηρητές από την Ευρωπαϊκή Ένωση που έκαναν και κάποια σχόλια. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υποστηρίξει την ενίσχυση των προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα προς την ευθυγράμμιση με τα διεθνή πρότυπα, ιδιαίτερα το, η ελευθερία έκφρασης και η ελευθερία συνάθρησης και να υπάρχει δυνατότητα να εκφραστούν όλες οι απόψεις. Πρέπει να πούμε στην ε, κυβέρνηση των Μαλδιβών να επαναλάβουν πόσο σημαντικό είναι το κράτο δικαίου, η ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη και ο χωρισμό ε, ο διαχωρισμό των διαφόρων εξουσιών. Ε, θέλουμε, θέλουν οι Μαλδίβε να συνεργαστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προκύψουν μια σειρά από συστάσει ε, των ομάδων εμπειρογνωμόνων, των αποστολών εμπειρογνωμόνων που έγινε το 2016. Η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση θέλει να συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλουμε να τροποποιήσουμε το νομοθετικό πλαίσιο στις Μαλδίβες, τις διαδικασίες και τις πρακτικές στο δικαστικό επίπεδο. Μια δεύτερη ομάδα πυρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να περιλαμβάνει και συμβουλές προς το Γενικό Εισαγγελέα ε, των Μαλδιβών. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συνεχίσει να πιέζει την κυβέρνηση των Μαλδιβών ε, να διατηρήσει το μορατόριο γύρω από τη θανατική ποινή, έτσι ώστε να προχωρήσουμε να κάνουμε ένα ακόμα βήμα προς την κατάργηση της θανατικής ποινής. Επίσης, πρέπει να προωθήσουμε την εκπροσώπηση, ε, την πολιτική των γυναικών, τον, την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών, ε, τη χειραφέτησή τους και τη μείωση της βίας κατά των γυναικών. Επίσης θα πρέπει να συνεχίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από κοινού με τις αρχές της Μαλδίβας, των Μαλδιβών ε, την προσπάθεια για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος. Αυτό περιλαμβάνει συνεργασία στα διεθνή φόρα και υποστήριξη της έγκρισης μακροπρόθεσμων στρατηγικών για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης οικονομίας που βασίζεται σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα γνωρίζετε ότι οι Μαλδίβες είναι επικεφαλής της συμμαχίας ε, των μικρών χωρών νήσων ε, και αυτός είναι, εδώ φαίνεται ο ρόλος, ο θετικός ρόλος που μπορούν να παίξουν οι Μαλδίβες στη διεθνή κοινότητα. Τέλος, ε, ασχολούμαστε και με το θέμα της ε, παράνομης αλίας, της αλίας IUU, τελειώνοντας πρόεδρε, πιστεύω ότι ως, μια, ως νεαρή δημοκρατία θα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις η χώρα αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο για να βοηθήσει να συνδράμει την, τις Μαλδίβες για να ξεπεράσουν τις προκλήσεις αυτές. Εφόσον δεν υπάρχει επίσημη συμφωνία, ε, ζητούμε πιο τακτικό πολιτικό διάλογο με τη χώρα αυτή και είμαστε διεθυμένοι να εμβαθύνουμε τις σχέσεις μας με τις Μαλδίβες και να ενθαρρύνουμε τις βελτιώσεις και όχι απλώς να δαχτυλοδείχνουμε. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κρίσλερ, για την εισαγωγή σας. Τέσσερις συνάδελφοι θα ήθελαν να πάρουν το λόγο. Peaceful. I will... Δεν ε, θα δώσω το λόγο σε άλλους. Ε, να έχουμε δηλαδή έναν γύρο ερωτήσεων και απαντήσεων. Δύο λεπτά ο καθένας προτείνω και κατόπιν ε, ο κύριος Κρίσλερ να κλείσει. Ο κύρι... Αρνόντα Ζαν, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μιλάω στο όνομα του κύριου Κούκαν, ο οποίος ήταν το 2014 επικεφαλής της αποστολής παρατηρητών. Να σας πω λοιπόν τι λέει. Παρακολουθώ. Παρακολουθώ τις εξελίξεις ε, στις Μαλδίβες ε, από την αποστολή του 2014 και μετά και σχεδιάζω να επισκεφτώ τις Μαλδίβες ε, εντός του έτους. Χαίρομαι που οι αρχές της χώρας έχουν δώσει το πράσινο φως για αυτήν την δεύτερη αποστολή. Σημαντικό είναι να έχουμε επικοδομητική συνεργασία όσον αφορά την τελική έκθεση και την εφαρμογή της. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό καθότι θα πραγματοποιηθούν εκλογές το 2018 στις Μαλδίβες. Προσβλέπω στην ε, καλή μας συνεργασία στον διάμεσο χρονικό διάστημα. το 2015 και μετά διαπιστώνουμε ότι υπάρχει δύσκολη κατάσταση όσον αφορά την άσκηση θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως είναι το δικαίωμα ε, του λόγου και το δικαίωμα του ε, συνεταιρίζεστε. Σημαντικό είναι να μπορεί να συμμετέχουν οι πολίτες στη δημοκρατική λειτουργία της χώρας και χρειάζεται να παρακολουθήσουμε στενά τις εξελίξεις στον τομέα αυτών. Ε, παραμένει η προβληματική κατάσταση όσον αφορά την ελευθερία των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Είδαμε εκφοβισμό των ε, δημοσιογράφων ε, και εντός του έτους. Ε, είδαμε τον θάνατο του Ιαμέν Νασίντ και γι' αυτό νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα επίκαιρη η σημερινή συζήτηση και πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση στις Μαλδίβες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Παντζέρη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Κρίσλερ που περιέγραψε καλά την κατάσταση των δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου της Μαλδίβης. Εγώ θέλω να υπογραμμίσω την επανεισαγωγή της θανατικής ποινή από πλευράς της κυβέρνησης μετά από 60 χρόνια μορατορίου και θέλω εκεί να επιμείνουμε. Ο Πρόεδρος ε, Ιαμέν τον Απρίλιο ε, ανακοίνωσε ότι θέλει να ξαναρχίσει τις εκτελέσεις. Η νομοθεσία των Μαλδιβών προβλέπει ε, την θανατική ποινή για την καταδίκη ακόμα και ανηλίκων. Οπότε θα πρέπει να στείλουμε ένα ξεκάθαρο και ισχυρό μήνυμα κατά αυτή της απόφασή σα ζητώ. Αν στις λιμένες δικές μας ε, ε, διατάξεις θα, πρέπει να, θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη και ένα μήνυμα το οποίο θα συνοδεύσει και μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης και προς όσους ως τουρίστες μεταβαίνουν στις Μαλδίβες θα ήταν χρήσιμο για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε τις ενέργειες των αρχών των Μαλτίβων. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Λόιζινγκ έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά... Μπορώ να μιλήσω γερμανικά? Ωραία. Όσον αφορά τις περαιτέρω δημοκρατικές εξελίξεις ε, μετά από τη συζήτηση που είχαμε μέλη της αντιπολίτευσης μου φαίνεται ότι είναι πολύ σημαντικό να εμποδίσουμε μέχρι τις επόμενες εκλογές και μετά φυσικά αλλά επίκαιρο είναι αυτή τη στιγμή να φροντίσουμε να μην ε, ε, πουν στη φυλακή ή δολοφονηθούν, για να το πω ακόμη πιο δραματικά, άλλα μέλη της ε, αντιπολίτευσης. Διότι αν γίνει αυτό, τότε δεν χρειάζεται καν να πραγματοποιήσουμε την αποστολή παρατηρητών στις εκλογές. Άκουσα τις περιγραφές περί έλλειψης δημοσιογραφικής ελευθερίας, αλλά νομίζω ότι αυτή η διατύπωση είναι υπερβολικά ήπια. Πρέπει να βρούμε τη σωστή ισορροπία ανάμεσα στο να παραμείνουμε σε επαφή και να ασκήσουμε πίεση. Αυτό συχνά είναι δύσκολο. Πώς μπορεί να γίνει αυτό λοιπόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Κατόπιν όσον αφορά την τρομοκρατία. Είπατε ότι η κυβέρνηση δίνει μεγάλη σημασία στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Ε, αναρωτιέμαι όμως ε, πώς ακριβώς ε, ορίζει την τρομοκρατία, διότι για παράδειγμα ο κύριος Έρτογκαν θεωρεί τις συνδικαλιστικές δραστηριότητες τρομοκρατία και βάζει τέτοιους ανθρώπους στη φυλακή. Όταν βλέπουμε πόσοι ε, ε, στρατολογούνται από τις Μαλδίβες ε, για το Ισλαμικό κράτος και πόσο μεγάλη είναι η αύξηση και όλα αυτό δεν ταιριάζει πάρα πολύ καλά με αυτό που λέει η κυβέρνηση. Τι μπορούμε λοιπόν να κάνουμε για το θέμα αυτό. Και ερώτηση προς τους συναδέλφους να ε, επιδιώξουμε νέο ψήφισμα στο Κοινοβούλιο, διότι ε, έχουν αλλάξει πολλά από το τελευταίο. Ευχαριστώ. Κυρία Λούζινγκ, ε, η κυρία Λάμπερτ από τους Πρασίνους. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Βρίσκομαι εδώ με την ιδιότητα της επικεφαλής της αποστολής που συμπεριλαμβάνει και τις Μαλδίβες. Όσον αφορά το ψήφισμα, νομίζω ότι ε, για να συντάξουμε ψήφισμα θα πρέπει να πιστεύουμε ότι θα έχει και αποτέλεσμα και δεν βλέπω να υπήρξε κάτι τέτοιο ε, στο προηγούμενο ψήφισμα. Εμένα με ενδιαφέρει το πώς αναπτύσσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις επαφές της με τις Μαλδίβες και ποιες είναι οι δυσκολίες, διότι έχουμε επαφή μέσω της πρεσβείας στη Σρι Λάγκα, αλλά συχνά είναι πολύ δύσκολο για τους πρέσβεις να ε, κάνουν δουλειά σε γειτονικέ χώρες, διότι πρέπει να αιτιολογούν και όλα τα αεροπορικά ταξίδια για τις συνομιλίες αυτές. Πιστεύετε ότι η ανάπτυξη διαλόγου με την ε, Σαουδική Αραβία είναι κάτι γενικότερο με τις Μαλδίβες ή είναι κάτι που ενδιαφέρει τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Τζιν Λάμπερτ. Τέσσερις συναδέλφους ακούσαμε, τέσσερις ερωτήσεις. Θα ήθελα να ακούσουμε τις απαντήσεις σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ενδιαφέρουσες ερωτήσεις σας. Στηρίζουμε την αποστολή του κυρίου Κούκαν, ε, την αποστολή που έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο. Βρισκόμαστε σε στενή επαφή μαζί του και θα στηρίξουμε την επίσκεψη αυτή. Συμφωνώ απολύτως με τη δήλωση του κυρίου Κουκάν και συνεργαζόμαστε στενά μαζί του. Όσον αφορά τη θανατική ποινή, Θα συμφωνήσω ότι είναι απαραίτητο να έχουμε πιο ισχυρή θέση για το θέμα αυτό. Η κυβέρνηση εδώ και αρκετό καιρό ανακοινώνει ότι θα ξαναρχίσει τις εκτελέσεις, ε, κάτι που δεν έχει συμβεί ακόμα, αλλά θα πρέπει να επιμείνουμε στο θέμα αυτό. Τέθηκε, βρισκόταν πολύ ψηλά στο θεματολόγιο όταν η, επικεφαλής, ε, όταν η αρχική ε, μάλλον όταν ο αρχηγός ε, της Αποστολής Ευρωπαϊκής Ένωσης επισκέφθηκε ε, τις Μαλδίβες τον προηγούμενο μήνα και ανέφερε ότι επί της αρχής απορρίπτουμε την ε, χρήση της αντική ποινή. Βρίσκω πολύ ενδιαφέρον και θα ήθελα να επισημάνω και απέναντι σε εσά ε, το θέμα ότι θα μπορούσαμε να ευαισθητοποιήσουμε τους τουρίστες στο θέμα αυτό. Αλλά θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα χειριστούμε το θέμα. προς την κυρία Λουίζινγκ. Είναι αλήθεια ότι ο διάλογος με την αντιπολίτευση είναι δύσκολος, πραγματοποιείται όμως. Συνομιλούμε με μέλη της κοινωνίας των πολιτών. Ακούμε αναφορές ε, σχετικά με το πόσο δύσκολο είναι για αυτούς ε, να ε, δραστηριοποιούνται. Αλλά είναι δύσκολο από τη μία να ενθαρρύνουμε την κυβέρνηση να δημιουργήσει συνθήκες ίσου ανταγωνισμού για όλους. Διότι ταυτόχρονα κάποια στοιχεία της κυβέρνησης, όπως ανέφερα και εγώ και άλλοι, υιοθετούν τη σαφή πολιτική να εξαφανίσουν μέλη της αντιπολίτευσης ώστε να μην είναι σε θέση να συμμετάσχουν στις επόμενες εκλογές. Στον διάλογό μας ε, θα πρέπει να επιμείνουμε πάρα πολύ στο θέμα αυτό. Να αναφέρουμε δηλαδή ποιε είναι οι προσδοκίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τι επόμενε κοινοβουλευτικέ εκλογέ, που κανονικά έχουν προγραμματιστεί για του χρόνου. Η τρομοκρατία αποτελεί προτεραιότητα στις πολιτικές της κυβέρνησης, αλλά και εμείς Έχουμε ζητήσει από την κυβέρνηση να μας δώσει καλύτερο ορισμό του τι ακριβώς εννοεί, ποιοι είναι τρομοκράτες κατά τη γνώμη της. Για παράδειγμα, θα θέλαμε κατάλογο των ανθρώπων που πιστεύουν ότι ανήκουν σε τρομοκρατικές ομάδες. Και ποιο είναι το χαρακτηριστικό που κάνει έναν πολίτη των Μαλδίβων τρομοκράτη. Δεν είναι πολύ σαφές αυτό και με τον ευρύ ορισμό που υπάρχει η νομοθεσία μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές διαφορετικές περιπτώσεις. Η παρέμβαση της Jean Lambert αντικατοπτρίζει το δίλημά μας όσον αφορά το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε αποτελεσματικές διπλωματικές σχέσεις με τις Μαλδίβες συνομιλούμε με την κυβέρνηση, δεν έχουμε εκπροσώπηση στην πρωτεύουσα, το οποίο μας δυσκολεύει, διότι δεν ε, έχουμε διάλογο σε τακτική βάση. Πολύ θα θέλαμε να έχουμε μόνιμη παρουσία στις Μαλδίβες για να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε όλες τις προκλήσεις, αλλά για λόγους δημοσιονομικούς μάλλον δεν είναι πολύ ρεαλιστικό αυτό αυτή τη στιγμή. Όσον αφορά τη Σαουδική Αραβία, αναπτύσσεται μια σχέση που έχει να κάνει ε, με το πόσο κοντά είναι οι κουλτούρες των δύο αυτών χωρών. Ε, υπάρχουν όμως και εμπορικά συμφέροντα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Thank you so much, Mr. for coming. Ευχαριστώ κύριε Κρίσλερ που ήρθατε στην ε, Επιτροπή μας. Νομίζω ότι ήταν πολύ σημαντική η ενημέρωση που μας δώσατε. Οι πολιτικές ομάδες θα πρέπει να αποφασίσουν, θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα υπάρξει νέο ψήφισμα ή όχι. Καλούμε λοιπόν τα κράτη-μέλη, καλούμε λοιπόν τις πολιτικές ομάδες να σκεφτούν αν κάτι τέτοιο θα είχε νόημα ή όχι. Περνάμε στο σημείο 4, έχουμε 15 λεπτά στη διάθεσή μας ακριβώς. Θέσπιση μηχανισμού συμβολής στη σταθερότητα και την ειρήνη. Εξέταση των τροπολογιών και περαιτέρω βήματα στην πολιτική διαδικασία. Πρόκειται για την τρίτη συζήτηση στην Επιτροπή μας ε, μετά από την συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, στις 21 Μαρτίου και την εξέταση της έκθεσης ε, στις 22 Μαΐου. 99 τροπολογίες υποβλήθηκαν μέχρι την προθεσμία της 8ης Μαΐου και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Αρνό Ντανζόν που είναι εισηγητής. Παρακαλώ. Président, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι αρκετά σύντομο γιατί έχουμε ήδη συζητήσει όπως θυμήσατε αυτό το κείμενο δύο φορές εδώ στην ε, αίθουσα αυτή και συζητήσαμε και με τους συναδέλφους των διαφορών ομάδων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις ομάδες που συμμετείχαν στη συζήτηση. Ε, όπως είχα πει όταν παρουσίασα αυτή την έκθεση, Πρόκειται για ένα τεχνικής φύσης κείμενο, καθώς πρόκειται για έναν κανονισμό. Πρόκειται δηλαδή για μια εργασία επί ενός νομικού κειμένου και κατά τη γνώμη μου η σημασία είναι να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε αυτό το κείμενο μέσα σε κάποιες λογικές ε, προθεσμίες χρονικές γιατί από αυτό εξαρτάται η αποτελεσματικότητα των αποστολών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δύσκολες περιοχές όπως το Μαλί, στην ε, Κεντρική Αφρική, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Ε, αυτά τα μέσα ακριβώς είναι μέσα που περιμένουν οι τρίτες χώρες που ε, όπου δρούν αυτές οι αποστολές και που χρειάζονται αυτή, αυτή την νομοθεσία. Πρόκειται για μια τεχνική λοιπόν εργασία που έπρεπε να γίνει ενός νομικού κειμένου. Η συζήτηση ωστόσο αποτέλεσε την ευκαιρία για μια πραγματική πολιτική φύση συζήτηση με πολύ σαφείς απόψεις που εκφράστηκαν. Ορισμένες ομάδες θεώρησαν εξ αρχής ότι η νομική βάση αυτού του κειμένου δεν ήταν εγγυημένη και άρα κράτησαν μια προσέγγιση διαφορετική από αυτή που εγώ είχα ε, επιλέξει, το σέβομαι αυτό. Άλλες ομάδες ακολούθησαν τις δικές μου συστάσεις και τους ευχαριστώ. Και έπειτα Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, πιστεύω, που ξεκίνησε με τους σοσιαλιστές για την πολιτική και δημοσιονομική διάσταση αυτού του μέσου. Και θα ήθελα να πω ότι σέβομαι απολύτως αυτή τη διάσταση. Πιστεύω πως πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το κείμενο επί το οποίο θα εκφραστούμε και θα ψηφίσουμε είναι κάτι το μεταβατικό, που θα καλύψει δηλαδή τα τρία επόμενα χρόνια. Και είναι αλήθεια ότι αρκετέ αντιρρήσει των συναδέλφων σοσιαλιστών αφορούν την ε, ε, βιωσιμότητα την ε, δημοσιονομική και την πολιτική αυτού του μέσου. Πιστεύω πως η συζήτηση θα έρθει. Κατανοώ την, ε, τον προβληματισμό αυτό, γιατί στο μέλλον το Συμβούλιο και η Κομισιόν, αν θέλουν αυτό το μέσο να συνεχιστεί, θα πρέπει να κάνουν νέες προτάσεις. Και πιστεύω πως από αυτή την άποψη οι αντιρρήσεις και οι παρατηρήσεις που διατυπώθηκαν θα έχουν ληφθεί υπόψη. Γι' αυτό και πρότεινα, και θα δούμε αν θα μπορέσουμε αυτό να το εφαρμόσουμε, μια συμβιβαστική διατύπωση ε, που θα μας επιτρέψει ταυτόχρονα να, εγκρίνουμε γρήγορα το κείμενο που έχουμε σήμερα μπροστά μας και να το διατηρήσουμε όσο γίνεται περισσότερο στην αρχική του μορφή που κατά τη γνώμη μου ε, προσφέρει κάποιες νομικές εγγυήσεις. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε και θα δούμε με ποια μορφή θα το κάνουμε αυτό, σημειώνοντας και ε, εδώ παραπέμπω στο αίτημα κάποιων ομάδων ότι τα χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν για αυτό το μέσο δεν θα πρέπει να προέλθουν από το μέσο ε, για τη συνεργασία και την ανάπτυξη. Και εδώ δεσμεύομαι να μπει στο συμβιβαστικό κείμενο που θα σας ε, προτείνω για υιοθέτηση. Σε αυτό το στάδιο βρισκόμαστε. Εάν τώρα δεν μπορέσουμε να περάσουμε το κείμενο και θα το συζητήσουμε στην επόμενη συνεδρία των συντονιστών. Έχουμε συμβαστικέ που θα καλύψουν τι περισσότερε από τι ε, τροπολογίε που έχουν υποβληθεί, αλλά βέβαια θα είναι πολύ πιο δύσκολο γιατί έχουμε ένα σωρό τροπολογίες με διάφορα σημεία τα οποία είναι δύσκολο να περάσουν. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Ερνό Ντονζό. Τρίτη ανταλλαγή απόψεων. Έχουμε μόνο 15 λεπτά, ωστόσο έχω αρκετούς συναδέλφους που θέλουν να πάρουν το λόγο. Mr. Vistisen, Ms. Wautmans, Ms. Lochbieler, Mr. Mrs. Lösing, and Mr. Carver. Okay, well, try and keep it as short as possible. At best would be a minute each. Λοιπόν, ένα λεπτό έκαστος. Ε, λοιπόν, ξεκινάμε τους κοιόδες. Πρώτος, Ο κύριος Κύριε Πρόεδρε. Παρακολούθησα συνεδρίαση των σκιωδών την οποία διοργάνωσε ο κύριος Δανζόν. Μία ήταν ε, ε, ε, η εξαίρεση του, αποκλεισμού του ECI και η άλλη ήταν για την ε, βιωσιμότητα. Πήρα τις, αυτές τις δύο τροπολογίες και τις συζητήσαμε. Είχαμε ομοφανία όσον αφορά τον αποκλεισμό του DCI και δύο διαφορετικές ιδέες για το πώς θα ενισχυθούν οι πτυχές αναπτυξιακής πολιτικής. Μία ε, Θα πρέπει να έχουμε ένα πιο συγκεκριμένο ορισμό όσον αφορά τους όρους, τους θετικούς ή τους αρνητικούς, ε, θετικές ή αρνητικούς καταλόγους για το ποιους σκοπούς θα μπορούν να υλοποιήσουν αυτά τα χρήματα. Έχω αύριο το πρωί καλέσει εκπρόσωπο της ΑΕΣ για να δώσει τη γνώμη της. Και στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να φτάσουμε σε μια συμβαστική λύση. Θα γίνει μια ψηφοφορία στην Επιτροπή ΔΕΒΕ την ερχόμενη Δευτέρα το απόγευμα. Αυτή είναι η κατάσταση. Δύο διαφορετικά μοντέλα λοιπόν για το πώς θα ενισχυθεί το, το σκέλος που αφορά τις ε, ε πολιτικές ανάπτυξης. Λοιπόν, πράγματος και ο εισηγητές πρώτα ο Μαμίκινς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, κάποιες συναντήσεις, ε, συζητήσεις έγιναν στην συνεδρίαση των ε, ε, σχεδόν εισηγητών. Όπως συχνά στο Κοινοβούλιο είχαμε διαφορετικές απόψεις. Οι εκπρόσωποι κάποιων πολιτικών ομάδων είπαν ότι οι ομάδες τους δεν πρόκειται να υποστηρίξουν αυτή την νομοθετική πρόταση. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι διατηρημένη να την υποστηρίξουν όμως. Είναι όμως απαραίτητο να συζητηθεί ε, να συζητηθούν κάποια σημαντικά στοιχεία. Πολλά μέλη τη δική μα πολιτική ομάδα, οι Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν συμφωνούν να χρησιμοποιηθούν χρήματα από τα κονδύλια ανάπτυξη για αυτό το εργαλείο. Δεν είναι πολλά τα χρήματα βέβαια, αλλά δεν μπορούμε να προβλέψουμε τι θα συμβεί στο μέλλον με τη χρηματοδότηση. Ελπίζω λοιπόν να υπάρξει υποστήριξη από του συναδέλφου για το θέμα αυτό. Ένα άλλο προβληματικό ζήτημα είναι τα κριτήρια για να υποβάλει κανεί ε, αίτηση για χρηματοδότηση. Ε, ο μηχανισμός για να αποφευθούν και οι παρανοήσεις όταν η πρόταση θα ψηφιστεί εδώ στο Κοινοβούλιο αλλά και στο μέλλον όταν το νέο αυτό εργαλείο θα αρχίσει να εφαρμόζεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Μαμίκινς και τώρα ο κύριος Βίστης και ο εισηγητής και αντιπρόεδρος μας. Ευχαριστώ τον ευχαριστώ τον εισηγητή για τη δουλειά που έχει κάνει, λέει ο κύριος Βίστησεν. Ε, εφόσον αυτό το εργαλείο αποδειχθεί αποτελεσματικό, πρέπει να δώσουμε ένα περιθώριο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Υπηρεσία Εξωτερική Δράση για να το εφαρμόσουν. Βεβαίω, αντιλαμβάνομαι τι ανησυχίε που ακούγονται για τη χρηματοδότηση, για το πώ θα προχωρήσουμε, πόσο μεγάλη θα είναι, θα είναι το πεδίο, πόσο μικρό. Ε, πρέπει όμω πρώτα να το χρησιμοποιήσουμε. Εάν δεν, το, δώσουμε αυτή τη δυνατότητα, ε, δεν ξέρω αν πρέπει να υπάρξει το εργαλείο γενικότερα. Εμεί θα το δούμε αυτό στην ομάδα μου, στην ECR. Ενδεχομένω να μπορέσουμε να το υποστηρίξουμε τελικά, διότι θεωρούμε ότι η αρχική ιδέα είναι καλή και η ιδέα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι καλή, εν πάση περιπτώσει, να του ε, δοκιμάσουμε για μια περίοδο και να το αξιολογήσουμε. Όμω, εάν αυτό τελικά προχωρήσει με τόσου περιορισμού και δικτύε ασφαλεία και δεν υπάρχει τελικά χρήση, ε, δεν ξέρω αν έχει νόημα έτσι το βλέπουμε εμείς και αυτό θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ε, και ε, στη συνεδρίαση με τον εισηγητή. Μάλιστα, επόμενο και ο εισηγητή είναι η κυρία Βάλτμαν από την Μαρτ Άλντε. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι πρώτα απ' όλα όπω και οι υπόλοιποι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή τον κύριο Λονζόν για την πολύ σκληρή δουλειά του σε αυτό το δύσκολο φάκελο. Εμείς συμφωνούμε με τον εισηγητή, τον υποστηρίζουμε. Έχει γίνει οικονομική προσπάθεια και από όλου του άλλου κύριου εισηγητέ και αυτό το εκτιμούμε. Και πολλά στοιχεία τη έκθεση τη ΔΕΒΕ, που μόλι τη ΔΕΒΕ λήφθησαν υπόψη, είναι αυτό το εργαλείο, αυτός ο μηχανισμό συμβολή σταθερότητα και στην ειρήνη θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιείται σε εξαιρετικέ περιπτώσει. Η πρόταση δίνει έμφαση στο γεγονό ότι η ανάπτυξη δεν είναι εφικτή χωρί ασφάλεια και ειρήνη και τούμπαλιν. Και εδώ παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο αυτή η διαδικασία. Συμφωνώ με την Κομισιόν και με τον εισηγητή ότι σε κάποιε ε, συνθήκε η υποστήριξη ε, η στρατιωτική είναι απαραίτητη. Τέλο, να πούμε ότι είμαστε υπέρ αυτή τη ιδέα, διότι ε, η υποστήριξη αυτή ελέγχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θέλουμε λοιπόν να συνεχιστεί, να συνεχιστεί η συζήτηση για το φάκελο αυτό και να μπορέσει να προχωρήσει η Κομισιόν στη δουλειά τη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και τώρα κυρία Λόζινγκ από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνούμε με την επιχειρηματολογία των σοσιαλδημοκρατών. Ωστόσο, εμείς ε, θα το ορίζαμε με πιο ευρύ τρόπο. Το θέμα δεν είναι μόνο η πόρια από την αναπτυξιακή βοήθεια, αλλά ε, έχει να κάνει με γενικά την χρήση πόρων από τον προϋπολογισμό για στρατιωτικούς σκοπούς. Και δεν καταλαβαίνω πώς ο εισηγητής μπορεί να λέει ότι βρισκόμαστε νομικά σε στέρεο έδαφος, διότι οι νομικοί έφτασαν στο συμπέρασμα ότι αυτή η πρόταση δεν συνάδει με τις συνθήκες. Η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου καθώς και η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου κατέληξαν ε, σε αυτό το συμπέρασμα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό λοιπόν. Τι, τελείωσε ο χρόνος μου. Α, καλά. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Λόχπίλερ από τους Πρασίνους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλώ στο όνομα της Εμπότιλ Βαλέρο που είναι σκιώδης η συγγήτριά μας και που δεν μπορεί να είναι παρούσα σήμερα. Σημειώνουμε, κύριε Ισηγητά, ότι έχετε αποσύρει όλες τις τροπολογίες σας και χωρίς επιφυλάξεις δέχεστε την πρόταση της Κομισιόν του Ιουλίου του 2016. Αυτή είναι μεγάλη στροφή και σας καλούμε να εξετάσετε μήπως ε, θα πρέπει να αμφισβητηθεί το σύνολο της πρότασης της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου η νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου στη γνωμοδότησή της του Αυγούστου του 2016 λέει ακριβώς αυτό. Το θέμα εδώ είναι να έχουμε κανόνες που να σέβονται την ε, ε, νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Και θέλουμε να υπερασπιστούμε όχι μόνο το μέσω αυτό της ε, άμυνας, ε, αλλά να σεβόμαστε και τους ισχύοντες κανόνες. Επίσης, ε, δεν παίρνουμε μόνο πόρους από την αναπτυξιακή βοήθεια. Είναι πολύ ευρύτερο το θέμα και μας απογοητεύει Πιστεύει πολύ το ότι δεν το βλέπετε αυτό. Ευχαριστώ, James Κάβαμ, από το EFTD. Σας ευχαριστώ, ε, κύριε Πρόεδρε. Ε, πρέπει να αμφισβητήσω το κατά πόσο είναι απαραίτητο η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει δράση στο θέμα αυτό. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί περίτο επίπεδο και ε, το όλο κίνητρο εδώ πέρα είναι οι φιλοδοξίες διαφόρων όσον αφορά την έκθεση αυτή. Ε, όπως ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι, έχουμε αμφιβολίες ε, όσον αφορά τον όρο Military Actor. Θα έπρεπε να είναι πολύ πιο σαφής η διατύπωση του εισηγητή. Κάτι που θα μπορούσε να ε, ανακουφιστεί πολλές από τις ανησυχίες των συναδέλφων είδαμε στη Μέση Ανατολή ε, όπου εξοπλισμός από τη Δύση επιδίνωσε την κατάσταση και ουσιαστικά ήταν περισσότερο η ζωάρος μας. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να απορρίψουμε την ε, διεύρυνση του ταμείου αυτού. Ευχαριστώ τον James Carver. Έχουμε άλλους δύο μιλητές από το S&T, ο Κνούτ Φλέκενστάιν και μετά η Άννα Παρακαλώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Αρνόντον Ζων για την ετοιμότητά του να βρεθεί συμβασμό. Εγώ νομίζω ότι είναι λογικά και απαραίτητα τα μέσα αυτά. Θα συνομιλήσουμε μαζί του σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής ΔΕΒΕ. Και τελικά η Επιτροπή ΑΦΕΤ θα αποφασίσει σε τι βαθμό μπορεί να εγκρίνει τη γνωμοδότηση υπάρχει πρόβλημα οικονομικό. Το δέχεστε αυτό. Και για να μην προδικάσουμε τις εξελίξεις για το μέλλον. Αλλά λέμε επίσης ότι άσχετα από αυτό, μετά την τριετία στο πλαίσιο της μεσοπρόθεσης ε, του μεσοπρόθεσμου οικονομικού προγραμματισμού θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει. Μαζί με τους συναδέλφους από την Γιούρη προσπαθούμε να καταλήξουμε σε κοινή προσέγγιση ώστε να είναι σαφές εγκαίρως πριν την ψηφοφορία αν υπάρχει πλειοψηφία υπέρ της πρότασης αυτής ή όχι. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Σας ευχαριστώ κύριε Φλέκερστάιν. Ε, ο κύριος Λίτς, σας ευχαριστώ πολύ για τις ε, συζητήσεις αυτές. Είναι απαραίτητες και γι' αυτό είναι και απαραίτητο να διαθέσουμε τον απαραίτητο χρόνο. Βλέπω, παίρνω πολύ στα σοβαρά τις ε, νομικές επιφυλάξεις που υπάρχουν. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό εδώ να μείνουν απ' έξω οι πόροι της αναπτυξιακής βοήθειας, του DCI, και θα πρέπει να δούμε τι συγκεκριμένα λέει η πρόταση αυτή. Υπάρχουν τέσσερα θέματα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να χρηματοδοτούνται. Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένας θετικός ή αρνητικός κατάλογος Ε, έχουμε και την γνωμοδότηση της Γιούρη. Θα δείξει συζήτηση προς τα που θα κηρυθούμε. Ευχαριστώ κύριε Λίτς. Να δώσω το λόγο στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ε, η κυρία Χάρτεμαν είναι παρούσα. Έχετε το λόγο αν θέλετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ισηγητά, Κύριοι Ευρωβουλευτέ, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την γενική του υποστήριξη προ την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τροποποιηθεί το μέσο συμβολή στη σταθερότητα και την ειρήνη και για τι προσπάθειέ του να βρεθεί συμβιβασμό. Εκτιμούμε τι προσπάθειε του κυρίου Ντανζάν να βρεθεί κοινό τόπο και τονίζουμε τον έκτακτο χαρακτήρα των προτινόμενων μέτρων. Πιστεύουμε ότι οι προσπάθειες του εισηγητή θα οδηγήσουν σε ικανοποιητικό αποτέλεσμα που θα επιτρέψει να προχωρήσει η διαδικασία. Προσβλέπουμε στην επικοδομητική συνεργασία στα επόμενα στάδια και προσβλέπουμε στην καλή συνεργασία με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για γρήγορη υιοθέτηση της πρότασης τροποποίησης του Μηχανισμού Συμβολής στη Σταθερότητα και την Ειρήνη. Και επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε να αναφερθώ σε τρία σημεία που αναφέρθηκαν κατά τη συζήτηση. Όσον αφορά τη σταθερότητα, θα ήθελα να πω ότι σκοπός της πρότασης αυτής είναι σε πραγματικά έκτακτες περιπτώσεις όπου ο στρατός να έχει να παίξει ρόλο κλειδί στην ε, καθιέρωση ή αποκατάσταση των συνθήκων που είναι απαραίτητες ε, για την σταθερότητα και θα ήθελα να αναφερθώ στο πλαίσιο που αναφέρεται στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και συγκεκριμένα τον στόχο υπαριθμών 16 που αναγνωρίζει τη σχέση ανάμεσα στην ασφάλεια και την ανάπτυξη με στόχο να προωθηθούν οι ειρηνικές ε, και ε, ε, ευημερούσες κοινωνίες. Τα κριτήρια λοιπόν ε, δεν επιτρέπουν ε, βοήθεια προς ε, τις στρατιωτικές δυνάμεις εκτός από πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου όπου ασχολούνται με την αναπτυξιακή βοήθεια. Και θα ήθελα να τονίσω ότι αυτή τη στιγμή το 88% σχεδόν το 90% της χρηματοδότησης ε, του Μηχανισμού Συμβολής στη Σταθερότητα και την Ειρήνη αναφέρεται ως επίσημη αναπτυξιακή βοήθεια και αυτή η τάση αναμένεται να συνεχιστεί. Λίγα λόγια επίσης όσον αφορά τους καταλόγους. Παρακαλώ να κλείσετε, λέει ο Πρόεδρος. Πολύ σύντομη παρατήρηση για τους καταλόγους. Ο σκοπός είναι να έχουμε μια σφαιρική προσέγγιση και οι συνάδελφοί μου που θα συνεργαστούν με τους ευρωβουλευτές ε, θα αναπτύξουν περαιτέρω το θέμα αυτό. Τέλος, όσον αφορά τη νομική βάση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τροποποίηση στον μηχανισμό συμβολής ε, στη σταθερότητα και την ανάπτυξη ε, και την ειρήνη με βάση τα άρθρα 209 και 212 της συνθήκης όπου μπορεί να επιδιωχθεί η αναπτυξιακή βοήθεια μέσω ενός ε, επιπλέον παράγοντα που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι στρατιωτικές δυνάμεις. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Χάρτεμαν. Φτάνουμε στις τελικές παρατηρήσεις του εισηγητή. Κύριε Ντονζόν, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ όλους όσους πήραν το λόγο. Θα ήθελα όλους τους ιδιαίτερους να ευχαριστήσω την ομάδα ALDE, ECR και τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτε, διότι είναι μια συζήτηση που δεν είναι και τόσο εύκολη. Πάντως υπήρξε βούληση για να βρεθεί μια επικοδομητική λύση με συμβαστικές λύσεις, συμβατικές, συμβαστικές προτάσεις. Ε, παραμένουν κάποια θέματα, όχι λεπτομέρειες βέβαια, κάποια ουσιαστικά ζητήματα τα οποία τον οποίο πρέπει να συμφωνήσουμε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε βέβαια ποτέ ποιο είναι ο τελικός στόχος. Αντιλαμβάνομαι κάποιε αντιρρήσει από άλλε πολιτικέ ομάδε, αλλά να θυμίσω ότι εδώ βιαζόμαστε. Μιλάμε για ένα κείμενο, ένα ε, εργαλείο το οποίο θα επηρεάσει την κατάσταση άμεσα, επιτόπου. Στι προηγούμενε δύο συζητήσει, εδώ έδωσα το παράδειγμα του Μαλή, όπου έχουμε αποστολές και στρατιωτικές ε, και μη στρατιωτικές που περιμένουν, περιμένουν ε, αγωνιωδώς να μπορέσουν να έχουν εξοπλισμό, ε, ιατρικό εξοπλισμό και στρατιωτικό, διοικητικό εξοπλισμό. Γι' αυτό εργαζόμαστε, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Αντιλαμβάνομαι βεβαίω κάποιες αντιρρήσεις νομικές, Ορισμένε φορές θεωρώ πάντως ότι υπήρχε και μια υπερβολή, διότι ορισμένε φορές η νομική ανάγνωση μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικά συμπεράσματα, τελείως διαφορετικά από αυτά που μας παρουσιάσαν οι πράσινοι, παραδείγματος χάρη. Τώρα για τη χρηματοδότηση και τον περίφημο κατάλογο των προϋποθέσεων, εντάξει, πρέπει να τα βρούμε αυτά, αλλά με καλή θέληση νομίζω θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Νταζό. Συνάδελφοι, να σας θυμίσω ότι θα συμβεί από εδώ και πέρα ψηφοφορία στην ΑΦΕΤ 11 Ιουλίου. Στη συνέχεια να σας πω ότι θα γίνουν δύο ψηφοφορίες. Πρώτα για την έκθεση, απλή πλειοψηφία και δεύτερη ψηφοφορία για την έναξη διαπραγματεύσεων όπου εκεί χρειάζονται 37 μέλη στους 73. Δηλαδή χρειάζεται υψηλή συμμετοχή και η Ολομέλεια, στην Ολομέλεια θα λάβει η χώρα ψηφοφορία του Σεπτέμβριο για την εντολή για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ και τώρα να περάσουμε στο σημείο 5. Ονομοδότηση της ΑΦΕΤ για την πρόταση δημιουργίας ενός συστήματος πληροφοριών και άδεια ταξιδίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορούμε να έχουμε στοιχεία από υπηκός τρίτων χωρών που δεν υπόκειται στην υποχρέωση θεωρήσεων από κοινού με τα διάφορα συστήματα και βάσει δεδομένων 154 τροπολογίες έχουν υποβληθεί, τα μέλη συμφώνησαν σε τρεις συμβαστικές λύσεις. Ο εισηγητής ή η εισηγητής, η κυρία Μπόντιλ Βαλέρο από τους Πράσινους, ενημέρωσε τη γραμματεία ότι δεν θα είναι παρούσα για την ανταλλαγή απόψεων. Ε, θα υπάρξει κάποιος που θα την καταστήσει. Ποιος θα την καταστήσει, η κυρία Λόχπίλερ, μάλιστα. Θα πρότεινα να δώσω το λόγο στην κυρία Λόχπίλερ πρώτα και στη συνέχεια θα ακούσουμε τους και Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Βαλέρο ευχαριστεί όλους τους συναδέλφους των άλλων πολιτικών ομάδων για την καλή συνεργασία. Παρότι η θέση των πρασίνων είναι θέση μειοψηφία στο θέμα αυτό. Το σύστημα πληροφοριών και άδεια ταξιδίου θα δίνει πληροφορίες για ταξιδιώτες που απαλλάσσονται από την υποχρέωση θεώρησης. Έτσι δίνονται εκ των προτέρων πληροφορίες, ε, πρέπει να συμπληρώνεται εκ των προτέρων ένα έντυπο και να δίνονται διάφορες πληροφορίες σχετικά με την ταυτότητά τους, σε κάτι που αντιστοιχεί ε, με ε, το σχετικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η γνωμοδότηση της ΑΦΕΤ περιορίζεται στα θέματα που έχουν να κάνουν με την εξωτερική πολιτική και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τρεις συμβαστικές προτάσεις υπάρχουν αυτή τη στιγμή και θα συνεχίσω στα αγγλικά για να μπω σε λεπτομέρειες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει αναθέσει μελέτη για να αξιολογηθεί ε, η σκοπιμότητα του αίτιας. Καταλήγει σε ένα συμπέρασμα που θα πρέπει να μας κάνει να ξανασκεφτούμε αυτά που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και να προσαρμόσουμε το ε, σύστημα. Ήδη έχουμε υπάρχοντα συστήματα όπως είναι το σύστημα πληροφόρησης Schengen και το νέο σύστημα ε, παραβιάζει τα ε, θεμελιώδη δικαιώματα. Γι' αυτό ε, η συγγήτρια αμφισβητεί την χρησιμότητα του αιτίας και πιστεύει ότι ο κανονισμός υπό τη μορφή που έχει δεν θα πρέπει να υιοθετηθεί. Η κυρία Βαλέρο υπέβαλε τροπολογίες που αναφέρονται στο στο άρθρο 29 για τα ύποπτα άτομα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη το σύστημα πληροφόρησης Schengen για να σταματήσει ε, την είσοδο πιθανών τρομοκρατών ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να έχουμε έναν νέο κατάλογο επιτήρησης αίτιας θα αποτελέσει επικάλυψη εργασιών, θα επιφέρει όμως και πιο ασαφή κριτήρια σχετικά με τους όρους υπό τους οποίους θα περιλαμβάνεται κάποιος στον κατάλογο. Δεν χρειαζόμαστε περισσότερα εργαλεία, χρειαζόμαστε τα απαραίτητα εργαλεία. Ο κατάλογος επιτήρησης ε, θα κάνει ε, θα προκαλέσει ακόμα περισσότερη σύγχυση. Θα ε, πλημμυρίσουμε από δεδομένα και έτσι πιθανότατα να γίνουμε λιγότερο ασφαλείς. Γι' αυτό θα είναι πιο καλό να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τις δυνατότητες των υπαρχόντων συστημάτων. Επιπλέον, το σύστημα ε, αναθεωρείται αυτή τη στιγμή και θα εισαχθούν ε, τροποποιήσεις πριν την υιοθέτηση του κανονισμού αίτιας. Έτσι θα μπορούσαμε να κάνουμε ακόμα πιο αποτελεσματικό το σύστημα αυτό χωρίς να δημιουργήσουμε πλέον, επιπλέον κατάλογο επιτήρησης. Έχουμε καταλήξει σε ε, συμβιβασμούς. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο φιλικό προς το χρήστη το σύστημα αίτιας και η πληροφοριακή εκστρατεία πριν την εισαγωγή του συστήματος θα πρέπει να υποστηριχθεί από τα κράτη-μέλη, πρεσβείες και αποστολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις εν λόγω Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον κύριο Πίλερ, και τώρα οι για το ΕΛΚ, ο κύριος Τέτινα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, ο κανονισμός αυτός αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα ε, για φέτος. Το ΕΛΚ υποστηρίζει την πρόταση. Για μένα το σύστημα αιτιάς θα είναι ένα από τα μέτρα το οποίο θα έρθει να αντισταθμίσει ε, την έλλειψη ελέγχων στα ιστορικά σύνορα του Σέγγεν. Στο παρελθόν υπήρχαν παρεμφερή συστήματα και στην Αυστραλία και στι ΗΠΑ και στον Καναδά. Πιστεύω λοιπόν ότι αυτό που λέει η Κομισιόν στην πρότασή τη ε, για την εισαγωγή με την εισαγωγή του αιτία ε, μειώνει ε, τον αριθμό ε, των αιτήσεων που θα δεν θα γίνονται αποδεκτέ, θα μειώνεται και η αναμονή στα σύνορα. Επίση θα αυξάνει την ασφάλειά μα και βελτιώνει τις δυνατότητες ταυτοποίησης προσώπων που ε, αποτελούν κίνδυνο. Θα ήθελα με τις τροπολογίες μου να απλοποιήσω ακόμα περισσότερο τις ε, διαδικασίες του αιτίας. Παραδείγματος χάρη πέρα από αυτά που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να υπάρχει δυνατότητα να υποβάλει κάποιος αίτηση ακόμα και σε κάποιο αεροδρόμιο, ακόμα και σε κάποιο λιμάνι ε, Αναμένω με ανυπομονησία την περαιτέρω συνεργασία με τον εισηγητή και του κοιόδη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Στέτινα και τώρα για, τους, για την ομάδα S&D ο κύριος Μπίνεφεϊ. Ευχαριστώ πρόεδρε και ευχαριστώ όλους για την εργασία τους. Πρόκειται για ένα μέτρο που γρήγορα θα προκαλέσει μεγάλες αλλαγές στη διαχείριση των εξωτερικών σύνορων της Ένωσης και στις σχέσεις με τις τρίτες χώρες. Από τη μια πλευρά μπορούμε να καταλάβουμε την προέλευση και την όλο ένα και πιο έντονη ε, ζήτηση από πλευρά των κρατών μελών της ενίσχυσης ε, των ε, συνόρων λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων. Από την άλλη πλευρά δεν μπορούμε να λάβουμε βεβαιασμένα τέτοιε αποφάσει, χωρί να σκεφτούμε ε, τις επιπτώσεις εις βάθος. Δεν είμαστε αντίθετοι στην αρχή μιας αυτόματης, ε, ενός συστήματος αυτομάτου ε, για έλεγχο των ταξιδιωτών προ την Ευρωπαϊκή Ένωση όπω υπάρχει στη ΣΥΠΑ και στον Καναδά. Όμω θα πρέπει να υπάρχουν κάποιε ασφαλιστικέ δεκλίδες. Όπω είπε και η συγκήτρια υπάρχουν διάφορε προτάσει από τι διάφορε πολιτικέ και έχουμε φτάσει σε κάποιες επιβαστικές. όσον αφορά την ομάδα μου. Εμείς προσπαθήσαμε να εστιαστούμε στην, σε εφαρμογές ε, των δικτύων εκτός της Ένωσης. Να εξηγήσουμε δηλαδή καλά ε, στις ε, χώρες όπου δεν προβλέπεται θεώρηση αυτά τα νέα μέτρα μέσω των πρεσβειών μας. Από την άλλη πλευρά θελήσαμε να εισάγουμε κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες για τους ετούντες ώστε να είναι πιο ασφαλής, ε, όσο γίνεται πιο ασφαλής η διαδικασία έγκρισης πέντε χρόνια δεν θα διατηρούνται τα ευαίσθητα στοιχεία πέρα από τη δυνατότητα σχηματισμού profiling, εάν υπάρχουν κάποιες, ε, κάποιοι προβληματισμοί ή υποψίες. Σε αυτό το σύστημα θα εφαρμοστεί για τα, εφαρμόζεται για τις χώρες ε, ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, αλλά και για τις χώρες όπως η Γεωργία ή η Ουκρανία που πρόσφατα απέκτησαν τη δυνατότητα χάρσης των θεωρήσεων ως αναγνώριση των προσπαθειών που καταβάλουν οι αρχές τους. Πρέπει να επιμείνουμε ε, ότι αν αυτό το σύστημα δεν, δεν είναι σωστά προετοιμασμένο θα εμποδίσει τους ταξιδιώτες, θα πρέπει να προσέξουμε τον αντίκτυπο το, στον τουρισμό και στις διπλωματικές σχέσεις της Ένωσης με τις τρίτες χώρες. Η πρόταση λοιπόν της Κομισιόν μπορεί να βελτιωθεί κατά τη γνώμη μου. Ευχαριστώ κυρία Μπότεμαν από τους φιλελεύθερους στην τελευταία ομιλήτρια. Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα να ευχαριστώ καταρχήν την κυρία Φαλέρο για το έργο της. Δεν είναι εδώ βέβαια, αλλά την ευχαριστώ παρόλα αυτά ε, για το ETIAS. Είναι μια πολύ καλή πρόταση. Είναι ένα ευρύ εργαλείο το οποίο αφορά τους υπηκούς των χωρών για να μην ε, ε μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι προσφέρουν κίνδυνο. Χωρί όπω η Αυστραλία, μέσα πολιτείε χρησιμοποιούν ήδη αυτήν την, ε, αυτό το σύστημα και επειδή θα αυξηθεί κατά 30% στο 2020 η κυκλοφορία, χρειαζόμαστε ένα εργαλείο το οποίο θα μας δίνει κάποιες πληροφορίες για αυτές τις εξαιρέσεις. Είμαστε λοιπόν ικανοποιημένοι με την πρόσθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όμως, ε, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να υπάρχουν οι απαραίτητες κλίδε ασφαλείας για να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που θα ε, τυχάνουν επεξεργασίας θα προστατεύονται και δεν θα χρησιμοποιούνται ε, με τρόπο μη ε, σωστό. Γι' αυτό υπάρχουν κάποιε δικέ ασφαλίσει και θεμελιώδη δικαιώματα. Ξέρετε, ε, ότι εμένα απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα των παιδιών, ε, των εξαφανισμένων παιδιών, των αγνοούμενων. Θα μπορούσε το αιτία να χρησιμοποιηθεί λοιπόν ω ένα εργαλείο για την εξέβρεσή του. Τώρα για τι τροπολογίε. Έχουμε φέρει μια τροπολογία για να φύγει η εκπαίδευση. Πολλέ ομάδε το έκαναν αυτό. Είναι σημαντικό να υπάρξει συμφωνία και από αυτού και όπω όλοι ξέρετε, πολλέ από τι συζητήσει για το φάκελο αυτό είχαν να κάνουν με το πότε που καταφέραμε να χρησιμοποιούμε το αιτία ε, για την παράτυπη μετανάστευση. Όπω ε, και σε άλλε ομάδε ε, υπάρχουν δύο απόψει. Σε κάποιου αρέσει, σε κάποιου δεν αρέσει. Εγώ προσωπικά είμαι υπέρ τη χρησιμοποίηση αυτού του εργαλείου και σε ό,τι αφορά την παράτυπη μετανάστευση. Όμω αυτό θα συζητηθεί κυρίω στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ Ελπίζω εκεί λοιπόν να βρεθεί μια λύση. Γιατί το γραμμές πάντως ε, σε ό,τι αφορά τις λίγες συμβαστικές λύσεις εμείς ε, συμφωνούμε. Ευχαριστώ. Θέλει κάποιος άλλος να προσθέσει κάτι. Όχι. Να σας θυμίσω ότι η ψηφοφορία στην ΑΦΕΤ θα γίνει στις 11 Ιουλίου. Και τώρα μπορούμε να περάσουμε στην πρώτη εξέταση δύο γνωμοδοτήσεων που έχουν να κάνουν με τη χρήση του συστήματος πληροφοριών Schengen είναι δύο γνωμοδοτήσεις ε, που είναι παρεμφερείς, οπότε θα έλεγα τα σημεία 6 και 7 να τα εξετάσουμε από κοινού. 37 τροπολογίε έχουν υποβληθεί για την ε, γνωμοδότηση σε διαφορετική χρήση του SIS στον τομέα των συνοριακών ελέγχων και 86 για την γνωμοδότηση σχετικά με τη χρήση του SIS για την επιστροφή των παράνομων διαμενών των υπηκόρων τρίτων χωρών χωρίς ε, περαιτέρω καθυστέρηση θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, την κυρία Χίλντε Βάντεμαν, να σας θυμίσω ότι έχουμε ακριβώς 15 λεπτά για να εξεταστεί το θέμα αυτό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Πάτε γρήγορα σήμερα, έτσι. Ε, με άλογο θα σας κυνηγάμε σε λίγο. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους και όλους τους για τη συνεργασία τους σε αυτήν την πέμπτη συνάντηση που έγινε την πέμπτη. Συμφωνήσαμε για τέσσερις προτάσεις συμβασμού ό,τι φορά για την, τη χρησιμοποίηση του ΣΥΣ για την επιστροφή ε, των, δια, των παράνομων και, άλλ, και άλλους τέσσερις για τους συνεργακούς ελέγχους. Γιατί η επίσημη συνεργασία η ανταλλαγή πληροφοριών, η διαχείριση των συνόρων, η, η διευκόλυνση των επιστροφών είναι σημαντικά στοιχεία. Το, το, χαρό, το παρόν σύστημα πληροφοριών σε λειτουργεί καλά, αλλά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ακόμα καλύτερα. Έτσι λοιπόν, καλωσορίζουμε τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είμαστε πεπισμένοι ότι οι αλλαγέ αυτέ θα ενισχύσουν τι δράσει τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα τη μετανάστευση και στον τομέα τη ασφάλεια. Οι συμβαστικέ πρωτοβουλίε με τι οποίε συμφωνήσαμε είναι περιορισμένε. Όπως γνωρίζετε, ένας, έχουμε μικρή αρμοδιότητα στο φάκελο αυτό ως ΑΦΕΤ, αλλά περιλαμβάνονται κάποια σημαντικά στοιχεία. Στους συμβασμούς και για τους δύο κεφακέλους επικεντρωνόμαστε στην κατάσταση των υπηκών τρίτων χωρών και των δικαιωμάτων τους. Παραδείγματο χάρη να εξασφαλίσουμε ε, τι θα γίνει με τις πληροφορίες που μεταφέρουν σε τρίτες χώρες. Ειδικέ εξασφαλίσεις για τους ε, ανηλίκους. Είναι η ηθική μας υποχρέωση ως μέλη της Επιτροπής ΑΦΕΤ να εξετάσουμε τα ζητήματα που αφορούν την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Όλοι θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι διεθνεί ασφαλεία οι σχετικέ είναι βασικέ αρχέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν θα πρέπει να το επαναλαμβάνουμε σε κάθε έγγραφο αυτό. Δυστυχώ όμω καθημερινά παραβιάζονται δικαιώματα επικών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό μα δείχνει πραγματικότητα. Πρέπει λοιπόν να έχουμε κατά νου ε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις χώρες μας ότι έχουμε κάποιες υποχρεώσεις απέναντι στους ανθρώπους. Και βεβαίως η κατάσταση είναι χειρότερη σε μη ευρωπαϊκές χώρες. Όμως αυτό δεν, αυτό δεν είναι λόγος η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην σέβεται, να μην προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα ίδια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξει ότι μπορεί να μοιράζεται πληροφορίες με πραγματικό τρόπο, σεβόμενοι όμως ε, τους δημοκρατικούς κανόνες και αξίες μας. Είμαι πεπισμένη ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε αυτό ε, νομίζω αποτυπώνεται στην ε, γνωμοδότηση και ελπίζουμε να μας υποστηρίξετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τώρα θα περάσουμε στους χειώδεις συγγητές. Έχει ζητήσει το λόγο η κυρία Σλούιτσα και ο κύριος Πίτσουλα. Η κυρία Λέζινγκ. μάλιστα. Λοιπόν, πρώτα ο κύριος Σίουτσα από την ΕΛΚ. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια, την κυρία Βάτμανς, για τη δουλειά της. Όπως γνωρίζετε, είναι ιδιαίτερα τεχνικά τα δύο θέματα αυτά, αφορούν κυρίως την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Έχουν προσθεθεί όμως διάφορες προτάσεις για να μπορούμε να ανταποκριθούμε ε, καλύτερα σε νέες ε, προκλήσεις ε, που σχετίζονται με την μετανάστευση και την ασφάλεια, που είναι μάλλον τα θέματα που συζητώνται περισσότερο αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο και θα συνεχίσουν να συζητώνται τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια. Πρόσφατα είχαμε την Παγκόσμια ημέρα προσφύγων και θα πρέπει να ανταποκριθούμε στις ευθύνε μας. Η περιοχή Σέγγεν και το σύστημα πληροφόρησης Σέγγεν ε, διασφαλίζουν τις βασικές ελευθερίες μας και στηρίζουμε ένα ισχυρό σύστημα πληροφόρησης Σέγγεν από πλευράς του ΕΛΚ. Είμαστε υπέρ της επικαιροποίησης του συστήματος ώστε να βελτιωθεί και να διασφαλίζει καλύτερα την ασφάλεια των πολιτών μας. Ωστόσο βρίσκω ότι η διατύπωση στις δύο γνωμοδοτήσεις ε, συχνά είναι υπερβολικά επικριτική και ε, υπονοεί ότι το σύστημα αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί καλά και παραβιάζει τα δικαιώματα. Ε, εμείς δεν συμμεριζόμαστε τη θέση αυτή. Πιστεύουμε ότι όσοι εργάζονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κάνουν εξαιρετική δουλειά σε ένα περιβάλλον γεμάτο προκλήσεις και θέλουμε ε, να συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους ανθρώπους αυτούς ε, με όποιο τρόπο μπορούμε. Γι' αυτό σήμερα έχουμε υποβάλει άλλη πρόταση στην εισηγήτρια για βελτιωμένη διατύπωση μιας από τις συμβαστικές τροπολογίες και βασιζόμαστε στη συνεργασία σας για να πετύχουμε ισορροπημένη λύση για όλους μας. Δεν έχει πάντα νόημα να προσθέτουμε ε, προτάσεις όπως με πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μεταναστών. Αυτές είναι βασικές αρχές ε, του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και η επανάληψη απλά οδηγεί σε πιο μακροσκελές και βαρύ κείμενο, κάτι που δεν κάνει πιο ασφαλή την περιοχή Σέγγεν. Όσον αφορά τον συμβιβασμό που λέει ότι τα παιδιά δεν πρέπει να αναγκάζονται να δίνουν δακτυλικά αποτυπώματα ή φωτογραφίε. Πιστεύουμε και πάλι ότι μπορεί να βρεθεί καλύτερη διατύπωση. Αυτό σχετίζεται με τι συμβαστικέ προτάσει 1 και 3. Ευχαριστούμε την κυρία Βάουτμανς και την γραμματεία της ΑΦΕΤ για όλη τη δουλειά που έχει γίνει και δηλώνουμε την ε, ετοιμότητά μας να συνεργαστούμε για να βρεθούν καλύτερες συμβαστικές προτάσεις για να βελτιώσουμε την ασφάλεια των πολιτών μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Σπίτσουλα. το σύστημα πληροφόρηση Σέγγεν η ραχοκοκαλιά το σύστημα πληροφόρησης ε, Σέγγεν είναι η ραχοκοκαλιά της ζώνης Σέγγεν και με τα νέα αυτά έγγραφα δεν δημιουργούμε νέο σύστημα, απλά βελτιώνουμε τη λειτουργία του παλιού συστήματος. Ε, βασικός στόχος είναι να βελτιώσουμε ε, την ε, λειτουργία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Ασφάλειας ε, και από πλευράς των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών έχουμε υποβάλει αρκετές τροπολογίες. Στο άρθρο 20 πιστεύουμε ότι σημαντικό είναι να τονίσουμε την συγκέντρωση δεδομένων διότι πρέπει να αναφέρεται και το όνομα του ατόμου και άλλα ονόματα που ενδεχομένως να έχει χρησιμοποιήσει ψευδόνυμα. Επίσης, Ε, στηρίζουμε την καλύτερη λειτουργία του συστήματος ε, πληροφόρησης ΣΕΝΙΕΝ και την ε, πιο αποτελεσματική εφαρμογή αποφάσεων και πιο αποτελεσματικές μεταναστευτικές ροές γενικά. Ωστόσο, ανοίγουν εδώ κάποια θέματα αρμοδιότητας, ιδιαίτερα εκεί που μιλάμε για ορισμό των συνόρων, διότι η Κροατία δεν έχει προσχωρήσει ακόμα στην ζώνη Σέγγεν και γι' αυτό δεν είναι πολύ σαφές το τι εννοούμε όταν μιλάμε για εξωτερικά σύνορα. Μιλάμε για εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξωτερικά σύνορα της περιοχής Σέγγεν. Γι' αυτό έχω υποβάλει τροπολογία για το άρθρο 12. Ε, σας ευχαριστώ. Ελπίζω μπορεί να μπορείτε να στηρίξετε την τροπολογία μου. Ευχαριστώ κύριε Πίτσουλα και η κυρία Λόιζινγκ από πλευρά της ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ. Μιλώ εκ μέρους του συνάδελφου ε, Μικελούρπαν που δεν μπορεί να είναι παρόν. Θα ήθελε καταρχάς ο συνάδελφος να ευχαριστήσει την εισηγήτρια. Θα στηρίξουμε οποιαδήποτε τροπολογία ε, βελτιώνει την προστασία των θεμελιωτών δικαιωμάτων. Παρότι είναι πολύ περιορισμένες οι αρμοδιότητές μας, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, τα δικαιώματα και η αξιοπρέπεια ε, του κάθε ανθρώπου να διασφαλίζεται. Και γι' αυτό είναι σημαντική για μας ε, η συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 4 όπου αναφέρονται τα προσωπικά δεδομένα και θα πρέπει να διασφαλίζονται τα δικαίωμα και πολιτών τρίτων χωρών που δεν βρίσκονται σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βασικό θέμα για μας είναι η διαβίβαση δεδομένων. Θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να μεταβιβάζονται δεδομένα ή βάσεις δεδομένων σε τρίτες χώρες ούτε σε περιπτώσεις επιστροφών. Καταδικάζουμε οποιαδήποτε ε, προσπάθεια να ε, συνδεθούν μεταξύ τους ε, η μετανάστευση με την εγκληματικότητα και την τρομοκρατία. Πιστεύουμε ότι το σύστημα το ευρωπαϊκό είναι τιμωρητικό και ότι αντίκειται στις ευρωπαϊκές αξίες μας. Είμαστε υπέρ όλων των τροπολογιών που προστατεύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ιδιαίτερα σε τρίτες χώρες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Λούιζινγκ. Να σας θυμίσω συνάδελφοι ότι η ψηφοφορία στην ΑΦΕΤ θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουλίου πάνω στα θέματα αυτά. Περνάμε τώρα στο σημείο 8 της ημερησίας διάταξης. Παρουσίαση της μελέτης η χρηματοδότηση του Ισλαμικού κράτους που ανέθεσε η Επιτροπή μας ε, μετά από απόφαση των συντονιστών. Η μελέτη αυτή εξετάζει τη φύση του Ισλαμικού κράτους και εξετάζει τους πόρους του και την οικονομική διαχείρισή του. Αναφέρεται και στις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας για να καταπολεμηθεί η χρηματοδότηση του Ισλαμικού κράτους. Ε, θα ήθελα να καλωσορίσω τον κύριο Jean-Claude Cousserin. Πού βρίσκεστε? και την κυρία Άγνες Λεβαλουά. Καλώς ήρθατε. Monsieur has been ambassador for France. Ο κύριος Κουσερόν έχει διατελέσει πρέσβης της Γαλλίας στην ε, Αιγύπτο, στην ε, Συρία και έχει επίσης διατελέσει ε, υπεύθυνο του Υπουργείου Εξωτερικών. Η κυρία Ντεβαλουά είναι ειδικό του σύγχρονου αραβικού κόσμου, είναι ερευνήτρια στην Διεθνή Ακαδημία Διπλωματίας και κατέχει την ε, θέση της Αντιπροέδρου του Ινστιτούτου Μελέτης ε, της ε, Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Επειδή έχουμε λίγο μείνει πίσω, δίχως άλλη καθυστέρηση, θα ήθελα να σας δώσω το λόγο ώστε να ενημερώσετε τα μέλη της Επιτροπής για τα κύρια πορίσματα αυτής της έκθεσης. Ποιος θα ήθελε να ξεκινήσει. Η κυρία, μάλιστα, η κυρία Ντεβαλουά. Και μετά ο κύριος Μπουσρό ίσως θα μπορούσατε να περιορίσετε τις εισηγήσεις στα 10 με 12 λεπτά ε, για να έχουμε κάποιο χρόνο για συζήτηση. Έχουμε 30 λεπτά για προβλέψη για αυτό το θέμα. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να σας παρουσιάσουμε αυτή τη μελέτη που έχουμε υλοποιήσει για τη χρηματοδότηση του ΝΤΑΕΣ, της Οργάνωσης Ισλαμικού Κράτος. Εγώ θα κάνω μια σύντομη εισήγηση και παρουσίαση για τα όσα γνωρίζουμε ε, για τη χρηματοδότηση αυτής της οργάνωσης και μετά θα δώσω το λόγο στον πρέσβη ε, Κουσρό. Το πρώτο σημαντικό σημείο που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι αυτή η οργάνωση Ισλαμικό κράτο, είναι σχετικά περίπλοκη και ότι είναι η πιο πλούσια τρομοκρατική οργάνωση στον κόσμο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε πώ λειτουργεί η χρηματοδότηση. Γιατί αυτή η οργάνωση είναι η πιο πλούσια στον κόσμο, γιατί είναι μια οργάνωση που έχει εγκατασταθεί σε μια επικράτεια με τη διαφορά από την Αλκάιντα που ήταν εκεί παρούσα πριν από τον ΤΑΕΣ εμπνέεται από αυτήν βέβαια τον ΤΑΕΣ, ωστόσο η μεγάλη διαφορά είναι ότι ελέγχει μια επικράτεια τέτοιο που το επιτρέπει να έχει στη διαθεσή του σημαντικούς οικονομικούς πόρους. Πρώτα απ' όλα το πετρέλαιο βεβαίως, γιατί η περιοχή όπου έχει κατασταθεί το ΤΑΕΣ ανάμεσα στη Συρία και το Ιράκ είναι μια ε, σημαντική πετρελαιακή ζώνη είναι μια επικράτεια επίσης που το επιτρέπει να ελέγχει φυσικούς πόρους όπως το βαμβάκι αλλά και το σιτάρι και υπάρχει και ολόκληρο το δίκτυο ε, λαθρεμπορίου, αρχαίο δίκτυο το οποίο επανενεργοποιήθηκε από αυτή την τρομοκρατική οργάνωση με συγκεκριμένα με ολόκληρη ε, λαθρεμπορία έργων τέχνης και αρχαιοτήτων γιατί όπως ξέρετε αυτή η περιοχή είναι το λίκνο της ανθρωπότητας με αρχαιολογία αρχαιολογικά αρχαιολογικούς χώρους ε, ε, τερα, και επίσης ε, μπόρεσαν να λελετήσουν τράπεζες και κυρίως την τράπεζα της Μοσούλης που επέτρεψε σε αυτή την οργάνωση να κάνει μια πρώτη σειρμαγιά 100 δις λέει η ομιλήτρια, δολαρίων που, του που τους επέτρεψαν να εγκαθριδηθούν στην περιοχή έπειτα. Φορολογούν την, τον πληθυσμό. Εφόσον λοιπόν το ΝΤΑΕΣ έχει εγκατασταθεί σε μια συγκεκριμένη επικράτεια, ελέγχει 8 εκατομμύρια κόσμο σε αυτήν την επικράτεια. Δηλαδή έχει εγκαταστηδρήσει ένα σύστημα εξαιρετικά σημαντικό φορολογίας και ε, αυτό τους επιτρέπει να μην χρειάζονται εξωτερική χρηματοδότηση, αλλά να έχουν αρκετούς πόρους με όλα αυτά τα στοιχεία που σας προανέφερα, ώστε να μπορούν να ζουν με αυτά τα χρήματα. Τώρα τι συμβαίνει. Έχουν ληφθεί φυσικά μέτρα για να σταματήσει η εδαφική επέκταση του ΝΤΑΕΣ και έτσι ώστε να μην μπορεί πλέον να έχει πρόσβαση σε αυτούς τους φυσικούς πόρους για τους σας μίλησαν και μίλησα και ε, γι' αυτό και βομβάρδισε ο Διεθνής, ε, η Διεθνή Συμμαχία ε, για να μην χρησιμοποιεί πλέον, να μπορεί, μην μπορεί πλέον να, να εκμεταλλευτεί τα πετρελαϊκά κοιτάσματα. Οι βομβαρδισμοί λοιπόν αυτοί επέτρεψαν την απώλεια πόρων γιατί έθεσαν εκτός λειτουργίας διάφορες ε, έθεσαν εκτός λειτουργίας τις πετρελοπηγές. Ε, περιορίστηκε δε και η επικράτεια την οποία ελέγχει τον ΤΑΕΣ. Τον ΤΑΕΣ αυτή τη στιγμή λοιπόν ε, πάει ε, πιο αργά, ε, έχει περιοριστεί στην χώρο που κατέχει από όταν ξεκίνησαν οι δραστηριότητες η δράση στο 2014 και έχει πολύ λιγότερου πόρου στη διάθεσή τη. έχει και λιγότερο κόσμο. Ε, άρα λιγότερα χρήματα μπορεί να πάρει από, το πλήθο, από τον πληθυσμούς που ελέγχει. Επίση, ο πληθυσμό αυτό έχει φτωχύνει ε, και άρα δεν μπορεί να έχει το έσοδα. Έχουμε λοιπόν μια οργάνωση που όπως είπα ε, χάνει ταχύτητα γιατί έχει πολύ λιγότερη χρηματοδότηση και άρα είναι και λιγότερο ελκυστική για τους νέους γιατί οι μισθοί που πρότειναν στην αρχή ήταν εξαιρετικά ελκυστικοί, είδαμε πολλούς νέους να φεύγουν ε, ε, και να στρατολογούνται γιατί τους πρότειναν μισθούς για τους μαχητές αλλά και ε, ελκυστικούς μισθούς ακόμα και για τους ε, οργανωτές και συντονιστές. Σήμερα δεν ισχύει πια αυτό. Να σας πω βέβαια ότι δεν σημαίνει πως έχει διαλυθεί η οργάνωση και ότι δεν έχει δυνατότητες να βλάψει. Ε, έχει όμως επίσης λάβει υπόψη το γεγονός ότι έχει λιγότερους πόρους στη διαθεσή της και έχει προσαρμοστεί σε αυτή τη νέα οικονομία που χρειάζεται να αντιμετωπίσει. Και είναι αλήθεια πως σήμερα έχει περισσότερες δυσκολίες να προσελκύσει μαχητές, γιατί όπως είπα δεν τους πληρώνει πια με τόσο ελκυστικούς μισθούς όπως στην αρχή και φαίνεται να υπάρχουν και εντάσεις ανάμεσα στους μαχητές γιατί εκτιμούν ότι δεν πληρώνονται όσο θα έπρεπε. Αντίθετα, αυτοί που ασχολούνται με την επικοινωνία για τον ΤΑΕΣ πληρώνονται περισσότερο αυτή τη στιγμή. η ΤΑΕΣ κατάλαβε ότι εφόσον έχει λιγότερους πόρους για να, για να ε, ελκύσει τους μαχητές, όφιλε να κάνει πολύ καλύτερη επικοινωνία, έτσι ώστε να φέρει κόσμο, να μπορέσει να ελκύσει κόσμο και νέους. Η οικονομία του ΝΤΑΕΣ λοιπόν έχει εξελιχθεί λόγω όλων αυτών των στοιχείων που σας ανέφερα εντάχει. Θα μπορούμε βέβαια να επανέλθουμε αν το επιθυμείτε. Και τελειώνοντας, γιατί νομίζω πως ε, έχουμε λίγο χρόνο, να πω μόνο ότι το ΝΤΑΕΣ δεν έχει πλέον τους ίδιους πόρους, ωστόσο εξακολουθεί να υπάρχει. Ε, αυτό πρέπει να είναι σαφές και ο πρέσβης ε, Κουσρών θα σας πει κάποια περισσότερα πράγματα για αυτό το δεύτερο στοιχείο. Agnès Η Ανιές Λεβαλουά μας εξήγησε πολύ καλά και ξεκάθαρα γιατί και πώς η οργάνωση αυτή έχει χάσει κάποιες από τις δυνατότητες της και πώς είναι οργανωμένη αυτή τη στιγμή. Έχει χάσει λοιπόν από την επικράτη, έχει χάσει από τους πόρους, έχει χάσει σημαντικούς, σημαντικά μέσα, αλλά και τον κεντρικό της χαρακτήρα και η οργάνωση είναι κεντρική σε σημαντικές πόλεις έχασε αυτές τις δυνατότητες, αλλά έχασε και πολλές δυνατότητες στήριξης και κυρίως είναι αντικείμενο όχι μόνο δράσης εξωτερικής, και ενό συνόλου μέτρων που έχουν λάβει διάφορες χώρες και που αποδυναμώνουν τις δυνατότητες της. Είναι αποδυναμωμένη η οργάνωση αυτή και έχει υποχρεωθεί να αλλάξει τη δομή της, την παρουσία της, τις φιλοδοξίες της και προσπαθεί να προσαρμοστεί. Όλοι οι παρατηρητές θεωρούν ότι αυτό δεν σημαίνει πως ε, έχει χάσει τις δυνατότητες της να δράσει και να βλάψει, ότι έχει χάσει τη δύναμή της. Όχι, οι περισσότεροι παρατηρητές θεωρούν ότι θα υπάρξει το μετά. Και αυτό πρέπει να σκεφτούμε. Ποιο είναι το μέλλον αυτής της οργάνωσης και του συστήματος χρηματοδότησης του, ε, της οργάνωσης και ποια μέσα θα εξακολουθεί να έχει στη διάθεσή της. Εδώ τα σενάρια δεν είναι γραμμένα. Πρέπει να σκεφτούμε και να δούμε ακριβώς ποιοι είναι οι παράγοντες που θα μπορούσαν σήμερα να αποκτήσουν σημασία για να μπορούμε να καταλάβουμε τι θα μπορούσε να συμβεί και πόσο και πώς θα μπορούσαν να βλάψουν από εδώ και μπρος, να βλάψει αυτή η οργάνωση. Πρώτα μια πρώτη υπόθεση που είναι αρκετά απλή και που ανέφερε και η Ανιές Λεβαλούα μπορεί αυτή η οργάνωση του ΔΕΣ να βγει από αυτό το σχήμα το εδαφικό, δηλαδή υπήρχε μια σειρά από κεντρικές οργανώσεις σε συγκεκριμένη επικράτεια, με πόλεις, πρωτεύουσα κτλ. Σήμερα όλα αυτά έχουν αλλάξει. Θα υπάρξει λοιπόν μια διάλυση, όχι μόνο μια αποδυνάμωση, αλλά και μια κατανομή διαφορετική. Δεν θα υπάρχει πλέον κέντρο. Με πώς θα γίνει ακριβώς αυτό δεν το γνωρίζουμε, αλλά ξέρουμε ότι μπορεί να καταφύγεται στο, σύστημα της ε, δημιουργίας θηγατρικών, όπως το κάνει και η Αλκάιντα σε μια πρώτη φάση, να προσπαθήσει να προσαρμόσει την οργάνωση, τη δυνατότητες ε, δράσης ε, στα νέα μέσα και δυνατότητες που θα έχει. Λέει θα στην, ε, κάποιοι λένε θα πάνε στην έρημο. Ε, θα το κάνουν όμως ή μήπως θα προσπαθήσουν να πάνε προς τις πόλεις και να δράσουν στις πόλεις. Μια έκφραση που χρησιμοποιείται από τον τύπο και που κατά τη γνώμη μου είναι ατυχής είναι η ιδέα μιας ε, low cost τρομοκρατίας. Πολύ κακή έκφραση. Ωστόσο θα επιλέξουν τρόπους δράσης που θα μπορούσαν να είναι λιγότερο δαπανηροί αλλά που δεν θα είναι λιγότερο επιθετικοί η δολοφονική, η επικίνδυνη. Υπάρχει λοιπόν ο κίνδυνος να υπάρξει να, να, να δοθεί έμφαση με επίκεντρο τα άτομα και όχι τις ομάδες σε πιο διασκορπισμένη δράση όπου η οργάνωση θα είναι πιο αποκεντρωμένη και με την διατήρηση ενός κεντρικού πυρήνα που θα συνεχίσει να οργανώνει της δράσης. Αυτή είναι μια ιδέα για μια πρώτη προσαρμογή της ΔΕΣ, που μπορεί όπως είπαμε να έχει λιγότερα μέσα και λιγότερες ανάγκες. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι στις, την 11η Σεπτεμβρίου, η 11η Σεπτεμβρίου μάλλον είχε κοστίσει σχετικά λίγα χρήματα ανά α, μέλος. Υπάρχει τρομοκρατία δηλαδή που είναι λιγότερο δαπανηρή που είναι το ίδιο επικίνδυνη αλλά όχι τόσο δαπανηρή. Η ευρωπαϊκή δράση μέχρι στιγμής ήταν ότι προσπαθήσαμε να κόψουμε τις ε, στρόφιγγες. Όμως ο οργάνωση είναι λιγότερο εξαρτημένη από τα χρήματα αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, αυτή η υπόθεση λιγότερο δαπανηρή και περισσότερο διασκορπισμένη είναι η μόνη. Όχι. Υπάρχουν και άλλα σενάρια. Αντίθετα, λέει, μία άλλη, αυτή η οργάνωση δεν θα δεχτεί αυτή την, τον διασκορπισμό και την απώλεια ουσία και θα προσπαθήσει να αξιοποιήσει αυτό που τη απομένει. Δηλαδή, η κεντρική οργάνωση που διασκορπίζεται μεν είναι ένα ένας μηχανισμός προπαγάνδας που λειτουργεί, μια δομή, μια οργάνωση που υπάρχει και που ίσως θα μειωθεί και πάλι μπορούμε να φανταστούμε και όπως είπα και πάλι εδώ δεν είναι βάσιμε αυτές τι υποθέσεις, είναι απλά σενάρια. Θα μπορούσε να δοθεί προτεραιότητα στην επιβίωση τη οργάνωση και τι δυνατότητε αναζήτησης νέων πόρων. Και πού θα αναζητήσει νέου πόρου, νέες τεχνολογίες, τεχνολογίε, το crowdfunding, την ιδέα τη ε, περαιτέρω χρήση, τη στήριξη που μπορεί να έχει, να κινητοποιήσει τη στήριξη που μπορεί να υπάρχει για εκείνη, αλλά και να χρησιμοποιήσει το λαθρεμπόριο διαφόρων ειδών. Έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί κάποιο είδο οικονομικές και κερδοσκοπικέ ε, λειτουργίες. Μπορεί να χρησιμοποιήσει σύγχρονες τεχνικές για να πολλαπλασιάσει τα μέσα χρηματοδότησης. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι υπάρχουν πολλές υποθέσεις για το μέλλον αυτής της οργάνωσης. Η μία χαμηλού κόστους, όπως είπαμε, διασκορπισμένες δράσεις ή δεύτερη ότι θα καταφύγει είτε στο λαθρεμπόριο είτε σε τεχνικές ε, ε, τύπου μαφίας για να προσπαθήσει να επιβιώσει. και να επιβιώσει η δομή λήψης αποφάσεων ε, όπως έχει σήμερα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λεβαλουά και κύριε Κουσερό. Και τώρα θα καλέσω τους συναδέλφους που το επιθυμούν να πάρουν το λόγο. Ένα συνάδελφος έχει ζητήσει. Ήθελα να δώσω πρώτα στον κύριο Κόρβεν Μίκε το λόγο, αυτό θα ήταν πολύ ιδιαίτερο, αλλά έχουμε από το ΕΛΚΑ, όχι, τους σοσιαλιστές, ο κύριος Πίτσουλα πρώτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα πολύ απλό ερώτημα θέλω να θέσω με τη χρηματοδότηση του Islamic State, του Ισλαμικού κράτους. Είναι προφανές ότι τα, χρώμα προέρχονται από τα, τα, τα χρήματα προέρχονται από τα εδάφη. Αλλά αυτή τη στιγμή χάνει τα εδάφη του ε, το Ισλαμικό κράτος. Τι γίνεται όμως με την διασυνοριακή χρηματοδότηση διεθνής χρηματοδότηση αναφέρω, ε, θέλω να πω, από το εξωτερικό, από χώρες του κόλπου ή και από αλλού, από την ξένη ενίσχυση. Μιλάμε συχνά για τους ε, ε, ε, ξένους μαχητές, αλλά τι γίνεται με την, με την ξένη ενίσχυση. Πού βρισκόμαστε όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Ναι, ευχαριστώ κύριο Σασεβίτσιους τώρα για τους ε, φιλελεύθερους. Ευχαριστώ πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και για την ενημέρωση σχετικά με αυτό το εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα, την χρηματοδότηση του ISIS δηλαδή. Ε, σε ποιο βαθμό είναι σαφές κατά πόσο έχουν γίνει προσπάθειες από άλλες οργανώσεις να μάθουν από το ISIS. είναι μια τεχνογνωσία που έχουν οι τρομοκράτες και θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτό και άλλες επικίνδυνες οργανώσεις παγκοσμίω, να χρησιμοποιήσουν δηλαδή στοιχεία από αυτά που ε, ε, αποτελεσματικά χρησιμοποίησε ο Άισις. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ από την ΚΟΕ, παρακαλώ Κόουσο, ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποιες πτυχές, οι οποίες δεν αναφέρονται και τόσο. Ε, λέτε βεβαίως αυτό που συμβαίνει, ότι αυτό που συμβαίνει στο Ιράκ είναι διαφορετικό από που συμβαίνει στη Συρία. Ε, βεβαίως υπάρχουν δυνάμεις του Ιρακινού ε, στρατού που βρίσκονται στο Ισλαμικό στρατό τώρα, στο Ιράκ, λόγω τουλάχιστον του κυρίου Μπρέμερ και δημιουργήθηκε και το, η κυβέρνηση σεχταριστική του κυρίου Αλμαλίκ ε, και βεβαίω είχαμε αυτά που είχαμε μετά στη Φαλούτζα και αλλού. Αλλά στη Συρία είναι διαφορετικά τα πράγματα. 89%, 89 ε, διαφορετικές εθνικότητες ε, ε, μαχητών έχουμε. Τώρα, τώρα για το λαθρεμπόριο πετρελαίου συζητήθηκε και στα ε, Ηνωμένα Έθνη. Ε, το, μιλάμε για το λαθρεμπόριο πετρελαίου στα σύνορα με την Τουρκία αλλά και το λαθρεμπόριο, το εμπόριο εργών τέχνης. Ε, είναι ενδιαφέρον εδώ από οικονομική πλευρά τι γίνεται. Εμφανίζονται τράπεζε στι χώρε του κόλπου, εμφανίζονται σε φορολογική παράδοση, παράδειση και στην Τουρκία. Δηλαδή παρότι χάνει το έδαφο, ε, αυτά τα δίκτυα ε, πρέπει να καταπολεμηθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, James Cover από την FTD, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Κόουσο είπε μερικά από αυτά που ήθελα να πω κι εγώ. Ε, υπάρχει κάποιο, κάποιο στοιχείο χρηματοδότησης ε, που να... Ε, Βεβαίω είναι αυτή τη στιγμή πληγωμένη η οργάνωση. Υπάρχουν όμως οικονομικά πολιτικά στοιχεία που να δείχνουν ότι ε, το Ισλαμικό κράτος ε, μετακινεί χρήματα Υπάρχουν ανησυχίες και για την Ιεμένη, όπως ξέρετε. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ό,τι αφορά αυτό που σημαίνει στην Ιεμένη. Πείτε μας την άποψή σας από αυτού. Ο κ. Κόβιν Μίκη έχει τώρα το λόγο, παρακαλώ. cokolwiek zupełnie, nie dowiedziałem się, ναι, έχω να κάνω δύο ερωτήσει. Ε, πρώτη, δεν γνωρίζω ποιο αγοράζει αυτό το πετρέλαιο. Όπω γνωρίζω, εγώ για παράδειγμα έχω συζητήσει εδώ με τον πρέσβη μια από τι χώρε τη Μέση Ανατολή που μου είπε πολύ ξεκάθαρα ότι οι αγοραστέ είναι Αμερικανοί. Έμαθα επίσης ότι η Τουρκία αγοράζει πετρέλαιο. Δεδομένων τη σημερινή της σημερινής τεχνολογικής μας εξέλιξης και δυνατοτήτων, πώς είναι δυνατόν να μην ε, ξέρουμε πού, πάνε, πού πάει το πετρέλαιο και γιατί δεν έχουν ε, βομβαρδιστεί οι πετρελοπηγές. Γιατί σε δύο μέρες θα μπορούσαν να καταστραφούν τελείως. Γιατί δεν έχουν καταστραφεί οι πετρελοπηγές και δεύτερο, το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω ίσως κάποιος να μην θέλει να τις καταστρέψει. Κάποιοι κερδίζουν από όλη αυτή την κατάσταση. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν αυτό το ερώτημα είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι αλήθεια, αλλά εγώ έχω ακούσει ότι το ΝΤΑΕΣ μεταφέρει τώρα τη δράση, τη δράση του στη Λιβύη. Αλλά δεν άκουσα τίποτα σχετικά με αυτό από εσά. Και τέταρτον, και οι δύο μιλητές πιστεύουν πως το ΝΤΑΕΣ θα επιβιώσει από τις επιθέσεις ε, του Αμερικανικού ε, συνασπισμού. Αλήθεια, θα πιστεύετε ότι θα επιβιώσει. Ο κύριος Σέμκε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Σέμκε. Σας ευχαριστώ για αυτές τις παρουσιάσεις που μας κάνατε, τις εισηγήσεις και για τη δυνατότητα που μας δίνετε να παρέμβουμε. Πρέπει να, παραδεχτώ ότι ούτε και εγώ κατάφερα να καταλάβω τελικά πώς γίνεται να συνεχίζει να έχει έσοδα από το πετρέλαιο ο, ε, από στατικής άποψη μπορεί πολύ εύκολα να εντοπιστούν ε, οι πετρελοπηγές που λειτουργούν. Γι' αυτό και δεν καταλαβαίνω πώς γίνεται εδώ και τόσα χρόνια χωρίς καμία α, πάυση να συνεχίζουν να λειτουργούν αυτές οι πετρελοπηγές. Δεύτερον, όπως λέτε, το ΝΤΑΕΣ φαίνεται να αποδυναμώνεται. Γιατί αποδυναμώνονται και μειώνονται και τα έσοδα της οργάνωσης. Όμως, θέλω να ρωτήσω, είμαστε πραγματικά σε θέση να ορίσουμε, να δούμε ποια είναι η κλίμακα της μείωσης αυτών των εσόδων. Γιατί, εάν χάνει πολλά, θα χρειαστεί εξωτερική χρηματοδότηση. Αυτό έχει αναλυθεί, γιατί κατά την άποψή μου αυτό θα ήταν ένα τρόπο να απομονωθεί από εξωτερικού πιθανού χρηματοδότε. Ευχαριστώ. Thank you, dear colleagues, for... Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι για τις ερωτήσεις σα. Θα πρότεινα 7 λεπτά συνολικά για να απαντήσετε. Δεν ξέρω πώς θα μοιράσετε το χρόνο μεταξύ σα, Ποιος θα ήθελε να ξεκινήσει. Πρώτα οι παρακαλώ. Σύντομα, για να απαντήσω στο σύνολο αυτών των ερωτήσεων, να σας πω ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι το ΝΤΑΕΣ έχει ακριβώς αυτό το ζήτημα της ε, εδαφική ε, ε, εδαφικής επικράτειας το γεγονός ότι μειώνεται η επικράτεια την οποία ελέγχει σημαίνει και μείωση των εσόδων αυτός είναι ο κύριος λόγος της μείωσης των πόρων του. Για το θέμα του πετρελαίου και τις απορίες που έχουμε, θα πρέπει να κατανοήσουμε πως το ΝΤΑΕΣ στις αρχές της ε, κατάστασή του στην, ε, στη χώρα αυτή χρησιμοποίησε τα δίκτυα λαθρεμπορίου που υπάρχουν ανέκαθεν σε αυτή την περιοχή. Φανταστείτε είναι μια έρημος αν δούμε τη ζώνη του Λάκα, της Λάκα που είναι η ε, πρωτεύουσα του ΝΤΑΕΣ στη Συρία. Ολόκληρη αυτή η περιοχή είναι ερημική με δίκτυα λαθρεμπορίου που υπάρχουν από πάντα. Και η οργάνωση αυτή είχε χρησιμοποιήσει για λογαριασμό της. Υπήρχαν ήδη δίκτυα και θηγατρικές Κάποιε φορέ έχουμε, δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε πώς είναι δυνατόν να οργανώθηκαν όλα αυτά. Μα τα δίκτυα υπήρχαν ανέκαθεν, είναι από αρχαιοτά των χρόνων, μέσα από το Ιράκ, μέσα από την Τουρκία, χωρίς απαραίτητο να έχει ληφθεί απόφαση από τα κράτη. Είναι αποφάσει των δικτύων αυτών που υπήρχαν ήδη, υπήρχαν ήδη εγκατεστημένοι εκεί. Και αυτούς εκμεταλλεύτηκε το Ίσις για να χρησιμοποιήσει και να ε, πλουτίσει από το λαθρεμπόριο. Τώρα, γιατί υπάρχει μείωση των εσόδων, γιατί έχουν ληφθεί ένα σωρό μέτρα για να δυσκολέψει αυτή η κατάσταση. Α πούμε, όσον αφορά το εμπόριο αρχαιοτήτων, υπήρχαν λαθρέμποροι που μπορούσαν ευκολότατα να τα πουλήσουν. Αυτή σήμερα δυσκολεύονται γιατί έχουμε φτιάξει συστήματα για να εντοπίζουμε αυτά τα, τα, τα ε, αρχαία ευρήματα, αλλά και για να δυσκολεύονται οι εμποροί να βρούνε αγοραστές. Δηλαδή κινήσεις παγκόσμιες, οι οποίες τελικά έχουν φέρει καρπούς. Δεν γκριζώθηκαν βέβαια τα, δίκτυα αυτά των λαθρεμπόρων, αλλά εν πάση περιπτώσει δυσκολεύονται περισσότερο να τα χρησιμοποιήσουν. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία. Και έπειτα, διεθνή χρηματοδότηση. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι ότι πριν να πάρει, να καταλάβει τη Φαλούτζα ή τη Μοσούλη, τον ΝΤΑΕΣ υπήρχαν διάφοροι ε, έμποροι, μεγαλοεπιχειρηματίε στο σύνολο τη περιοχή του Περσικού Κόλπου, αλλά όχι μόνο εκεί, που χρηματοδοτούσαν αυτέ τι ταξιαρχίε που δεν ήταν αρχικά του ΤΑΕΣ και του, ή του ε, ε, αλλά πολύ γρήγορα όταν όλοι αυτοί καταλάβανε την ιδεολογία και το τι ήθελαν να κάνει τον ΤΑΕΣ, κόψαν την χρηματοδότηση. Διότι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι έμποροι, οι επιχειρηματίες κατάλαβαν την απίθανη δυνατότητα, ε, ε, ε τις βλάβης που μπορούσαν να προκαλέσουν αυτοί. Αλλά παλιότερα, επειδή υπάρχει και μέσα στην ε, μουσουλμανική θρησκεία ε, το ζακάτ, δηλαδή αυτό που είναι υποχρέωση των μουσουλμάνων να μοιράζονται με την κοινότητά τους στην υπόλοιπη τα ε, παραπανήσια τους πλούτη, ε, το έκαναν χωρίς να έχουν καταλάβει ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Εγώ μόλις όμως το κατάλαβαν ότι δεν πρόκειται για φιλανθρωπικές οργανώσεις, γιατί αρχικά το ίσως έτσι παρουσιάστηκε ως φιλανθρωπική οργάνωση δήθεν. Κατάλαβαν ότι δεν έπρεπε λοιπόν πια να τους δίνουν χρήματα και ότι έπρεπε να πάψουν αυτή τη δήθεν φιλανθρωπική δράση. Απάντησε στα περισσότερα ερωτήματα η Αγγλική του Λαλουά. Να προσθέσω και εγώ ένα-δύο στοιχεία. Είναι αλήθεια, είναι σαφέ ότι το ΝΤΑΕΣ δεν τη φτάνει ε, ξαφνικά μία ε, ωραία πρωία σε ένα παρθένο περιβάλλον. Υπάρχουν ήδη προβλήματα εκεί, υπάρχουν, υπάρχει ήδη λαθρεμπόριο, τα σύνορα είναι χαλαρά, υπάρχουν πολλά, υπάρχει λαθρεμπόριο μεταξύ Ιράκ και Ιράν, μεταξύ Ιράκ και Συρία, μεταξύ Ιράκ και Τουρκίας. Αυτά είναι αποτελούν πραγματικότητα, οικονομική, κοινωνική. και από τον ίδιο τρόπο όλα αυτά τα εμπόρια δεν συνδέονται με την τρομοκρατία. Υπάρχουν μια σειρά από δίκτυα κοινωνικά, φιλετικά, ε, Υπάρχει και η κατάσταση των Σουνιτών, που στις περιοχές αυτές δυσκολεύονται ιδιαίτερα και κατά κάποιο τρόπο αυτή τη στιγμή είναι αποδυναμωμένες. Βρίσκονται σε μια κατάσταση δηλαδή που θεωρούν, θεωρούν ότι αδικούνται, ότι μειονεκτούν. Αυτά τα λαθρεμπόρια λοιπόν υπάρχουν και είναι δύσκολο να καταπολεμηθούν και προϋπήρχαν Αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις ή παρατηρήσεις. Παρακαλώ. Well, okay, well, we need, I've heard we're supposed to get a short presentation. Uh, Άκουσα ότι θα ακούσουμε μία σύντομη παρουσίαση. Προλαβαίνουμε μέσα σε πέντε λεπτά. Πέντε λεπτά το πολύ, παρακαλώ. Κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, καλημέρα σα. Παρουσιάσω εν συντομία μια μελέτη που έγινε με βάση ε, τι εικόνε του δορυφόρου του Κοπέρνικου κατά τη διάρκεια της περίοδου Φεβρουάριο του 2017 που θα μας δείχνει τη δραστηριότητα των ε, πετρελαϊκών εγκαταστάσεων Αυτά τα στοιχεία μας επιτρέπουν να δούμε ποια είναι η θερμική δραστηριότητα στα κεντρικά και στα ανατολικά της Ευρώπης. Αυτά τα διασταυρώνουμε με το που βρίσκονται οι πετρελοπηγές και αυτό μας επιτρέπει να δούμε ποια είναι η δραστηριότητα στα διάφορα σε διάφορε καταστάσει. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν δύο πετρελαϊκέ καταστάσεις που είναι δραστηριότητα και μία ε, εγκατάσταση ε, επεξεργασία πετρελαίου. Ε, δηληστήρια δηλαδή. Βλέπουμε εδώ δυτικά της Παλμύρας, στο κέντρο της χώρας υπάρχει μια εγκατασταση ε επεξεργασια πετρελαιου ε δηληστηρια δηλαδη βλεπουμε πυκνότητα, μια πυκνότητα θερμική που δείχνει ότι υπάρχει μεγάλη δραστηριότητα και αυτό επιβεβαιώνεται και από τα δεδομένα του Sentinel-2 εδώ με τις υπεριόδες ακτίνες βλέπετε λοιπόν εδώ το φυσικό αέριο που καίγεται. Ε, οι εικόνες αυτές μας επέτρεψαν να δούμε και πού λαμβάνει η χώρα, ε, πού λειτουργούν τα διαλυστήρια τα ε, κάπως ε, πρόχειρα. Βλέπετε εδώ τις δύο ζώνες. Βλέπετε εδώ δύο προπετάσματα καπνού, αριστερά και δεξιά και επίσης είναι εμφανές ότι, εδώ υπάρχει δραστηριότητα δηληστηρίων τα οποία όμως είναι πρόχειρα. Εδώ έχετε μια συνολική εικόνα των εγκαταστάσεων δηληστηρίων στην χώρα και των σταθερών μονάδων με τα πράσινα είναι τα ενεργά και κόκκινα, ε, τα κόκκινα είναι ε, τα, πρόχειρα. Εάν δείτε το Φεβρουάριο του 2017 λοιπόν εδώ στα γκρι είναι αυτά τα οποία έχουν στα χέρια τους ε, το ΝΤΑΕΣ με πράσινο ε, οι ε, δυνάμεις των ανταρτών, με κόκκινο οι στρατιωτικές δυνάμεις και με κίτρινο οι Κούρδοι. Βλέπετε λοιπόν το ΝΤΑΕΣ και οι Κούρδοι έχουν κυρίως αυτά τα πρόχειρα δηληστήρια και τα, και τα οι κυβερνητικές δυνάμεις έχουν κυρίως τις μόνιμες εγκαταστάσεις. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Okay, thank you. Ladies, or ladies. Μάλιστα, ευχαριστώ για τις παρουσιάσεις. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας συστήσω να ρίξετε μια πιο προσεκτική ματιά στην ανάλυση που μας παρουσίασε εδώ η πολιτική μας μονάδα, ε, ευχαριστούμε πολύ και τώρα θα περάσουμε στο σημείο 9. Πριν ξεκινήσουμε, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι το σημείο αυτό θα συζητηθεί και κλεισμένο το θυρών, μόνο δηλαδή ε, τα, τα, τα, τα, μέλη, οι μόνιμοι υπάλληλοι και το πολιτικό προσωπικό μπορούν να παραμείνουν, οι υπόλοιποι παρακαλώ να αποχωρήσουν.